Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα ο κύριος Ντοζόν και εγώ θα συμπροεδρεύσουμε για την σημερινή συνεδρίαση που έχει σαν θέμα την σημερινή κατάσταση, την επικαιρότητα στην κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Όλοι ξέρουμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση εκεί και τη Δευτέρα μας έγινε μια πολύ ενημερωμένη παρουσίαση που αφορά βεβαίως την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή. Πρόκειται για ταραχές που έχουν και θρησκευτικό και χαρακτήρα. Υπάρχουν αιτίες λοιπόν και θρησκευτικές ε, και εθνικές που έχουν οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τη Δευτέρα αναφέρει ότι θα πρέπει να οργανωθεί με μεγάλη ταχύτητα μια νέα επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά είναι πολύ ενδιαφέρον ε, η δική μας Επιτροπή από κοινού με τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας να έχουμε καταρχήν μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί, να δούμε πώς μπορεί να οργανωθεί με ταχύτητα αυτή η επιχείρηση. Έχουμε, όπως ξέρετε, και άλλη εμπειρία όσον αφορά την ταχύτητα των αποφάσεων του Συμβουλίου και εδώ σκέφτομαι την επιχείρηση στο Μάλι. Θα πρέπει με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο γρήγορα να μάθουμε να αντιδρούμε γιατί πραγματικά είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να εγγυηθούμε περισσότερη ασφάλεια για τους ανθρώπους επιτόπου. Υπάρχει βεβαίως και η πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει εκεί. Αυτό σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο μέχρι να φτάσουμε σε μία πραγματική σταθερότητα από πολιτικής απόψεως. Με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα εδώ πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει για την σταθεροποίηση και την ειρήνευση αυτών των περιοχών της Αφρικής, τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι περιφερειακές δυνάμεις, τι προετοιμασία φυσικά μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε θα έχουμε και την συνάντηση κορυφής με τις Ηνωμένε Πολιτείε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα θα μπορούσε αυτή η συνάντηση κορυφής να παίξει ένα ρόλο επικοδομητικό γενικότερα για την προετοιμασία κάποιων επιχειρήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Έλμαρ. Νομίζω ότι κάλυψες όλα τα σημεία. Έχουμε εδώ ένα πάνελ πολύ αντιπροσωπευτικό. Ο κύριος Βέσκοτ, ο κύριος Λενουάρ, εκ μέρους της ε, CSPD, αλλά και ο ταξίαρχος Κλαβέ, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γαλλία στο ΝΑΤΟ. Και φυσικά έχουμε και αρκετό χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την κατάσταση. Ο Έλμαρ μας ε, θύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και με το πρόσφατο Συμβούλιο και τα συμπεράσματά του έχει δεσμευθεί όσον αφορά αυτήν την επιχείρηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι όχι απλώς να ακούσουμε τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας, είναι πολύ ενδιαφέρον για μας να δούμε πώς λαμβάνει η χώρα αυτός ο σχεδιασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που το γνωρίζουμε. Πολλές φορές ακούμε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται πολύ μακριά σε τόπο και χρόνο από την πραγματική κατάσταση. Ο κύριος Λενουάρ λοιπόν θα μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα και ελπίζω να ακούσουμε και κάποια πράγματα για τις ομάδες μάχης, τα περίφημα battle groups, τα οποία συζητήθηκαν τον Νοέμβριο και που φυσικά δεν οδήγησαν σε αποτελεσματική απόφαση όσον αφορά τουλάχιστον την κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Θα δέσω το λόγο και στην κυρία Κρετού που σήμερα είναι εδώ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Φυσικά και η αναπτυξιακή διάσταση όλων αυτών των επιχειρήσεων στην Αφρική είναι μία πάρα πολύ σημαντική συνιστόσα. Η ασφάλεια είναι, αν θέλετε, δύο πυλώνες τους οποίους θα πρέπει να συνυπολογίζουμε στην Αφρική. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ε, καλημέρα σας κύριε Μπρόκ. Ευχαριστούμε κύριε Ντανζά που οργανώσατε αυτή την τόσο σημαντική ανταλλαγή απόψεων μαζί με εμά την Επιτροπή για την Ανάπτυξη που μας ενδιαφέρει προφανώς τόσο πολύ το θέμα αυτό. Είναι ατυχές που η Ευρώπη με την εξαίρεση της Γαλλίας ίσως συνολικά τουλάχιστον δεν έχει δώσει περισσότερη προσοχή τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Μια χώρα που είναι από τις φτωχότερες, τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πλέον ευάλωτες από την άποψη των κυβερνητικών ε, οργανισμών και των ε, δυνατοτήτων τη μετά την κρίση στο Μάλι, αντιμετωπίζουμε πλέον το γεγονό ότι τα πράγματα πολύ γρήγορα μπορεί να κλιμακωθούν. Η κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία ήταν πολύ δυσχερή επί πολλά χρόνια και υπάρχει μια ιδρική υποβάθμιση της των κυβερνητικών δομών και της οικονομίας. Οι ανθρωπιστικές συνέπειες της κρίσης ήδη φάνηκαν αυτή την εβδομάδα, όμως να θυμίσω ότι μιλάμε για μια χώρα με φοβερά αδύναμες ε, υποδομές. Μιλάμε για 900.000 εσωτερικώς εκτοπισμένους, το 1 τρίτο του πληθυσμού δηλαδή της χώρας. Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής μας τη Δευτέρα υπογραμμίστηκε ότι 8 τουλάχιστον φορείς ζήτησαν έκτακτη στρατιωτική επέμβαση για να ε, σταματήσουν οι ανθρωπιστικές αυτές ε, πιέσεις που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι σε γενοκτονία. Από την αρχή της εβδομάδας είδαμε κάποια πρώτα θετικά βήματα, με λόγια τη συμφωνία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, για την ε, αποστολή της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, και το θέμα είναι στην πράξη πώς ε, περισσότερου άντρε θα μπορέσουμε να κυκλώσουμε εκεί, να αποστείλουμε εκεί. Έπειτα η διεθνή κοινότητα δεσμεύτηκε 360 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων καταλαβαίνω ότι το 150 μόλις θα αφοσιωθούν ε, σε ανθρωπιστικούς σκοπούς, ενώ τουλάχιστον 80 για την ευρύτερη σταθεροποίηση, ανάπτυξη υπηρεσιών, υποδομών, ενώ πρέπει να πούμε ότι τα 360 εκατομμύρια είναι διπλάσια τουλάχιστον από όσα το ε, πρόγραμμα ανάπτυξη, το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη είχε, αφιερώσει στην χώρα, είχε αφιερώσει στη χώρα αυτή για το διάστημα 2008-2013. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αμελήσουμε. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ήταν ευάλωτη, ήταν ένα αποτυχημένο κράτος και είχε εντοπιστεί τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη του 2009 όταν ε, γινόταν λόγος για τα ευάλωτα κράτη στην Αφρική. Υπόθηκε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αντιμετωπίσει τις ε, δυσκολίες των κρατών που είναι ευάλωτα ήδη. Υπάρχουν κάποιε προσπάθειε τα τελευταία χρόνια και ελπίζω σήμερα το πρωί να ακούσουμε τι μπορεί να γίνει του ερχόμενου μήνε. Κυρίω όμω τι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια, πιο μακροπρόθεσμα, ώστε να ξεπεράσουμε τον ευάλωτο χαρακτήρα του κράτου αυτού. Θα χρειαστεί αφοπλισμός των ένοπλων παραστατικών ομάδων και να δούμε τι εμπειρίες μπορούμε να αντλήσουμε από τη μέχρι τώρα ε, προσπάθειά μας για να προχωρήσουμε. Η εκλογή της κυρίας Κατρίνης Σαμπαπάντσα ήταν ε, μια πολύ ενθαρρυντική ε, τροπή στα πράγματα, με θετικέ αντιδράσεις και στη χώρα της αλλά και με πρώτε δικές της θετικέ δηλώσεις. Ελπίζουμε ότι θα γίνει ένας πραγματικό μας εταίρος. ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ε, merci bien. Ευχαριστούμε. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του ταξιάρχου Κλαβές, του στατικού Κλαβές, για την ε, κατάσταση της ασφάλειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις από την πλευρά της Γαλλίας, ήδη από το Δεκέμβριο, με μια εντολή βεβαίως που είχε ανατεθεί από τον ΟΗΕ, και μετά θα ακούσουμε τον Διδιέ Λενουάρ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα με καλέσατε εδώ και θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ανταλλαγή Απόψεων θα σας παρουσιάσω βεβαίως την γαλλική άποψη. Δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει κανείς τα πάντα σε ένα τέταρτο. Όπως ξέρετε κάθε μέρα γίνονται έκτροπα, υπάρχει βία και ταραχές. Το να μπορέσει κανείς λοιπόν να σας ε, παρουσιάσει την κατάσταση, πώς έχει αυτή τη στιγμή, ε, δεν θα μας επιτρέψει να στραφούμε προς το μέλλον. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε τι είναι ανισχυτικό και τι είναι λίγο πιο ενθαρρυντικό. Θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία, κάποιες, ε, κάποια δεδομένα. Βεβαίω ο καθένα μπορεί να εκτιμήσει τελείω διαφορετικά την κατάσταση. Εγώ θα ήθελα και από στρατιωτική απόψεω να σας παρουσιάσω κάποια πράγματα που ενδεχομένω θα έχουν ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω λοιπόν παρουσιάζοντάς σας όπως το έχω προετοιμάσει το κείμενό μου. Καταρχήν οι εμπλεκόμενοι οι δυνάμεις που βρίσκονται επί τόπου, η Μίσκα και οι Σάγκαρες, οι δύο επιχειρήσεις, η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια, η ανθρωπιστική κατάσταση και βεβαίως θα αφήσω στο τέλος τον Διδιέ να μιλήσει για την διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά ειδικότερα την επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτόπου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις δυνάμεις, τις απειλές. Καταρχήν η εξ σελέκα. Είναι περίπου 6 με 8.000 άτομα. Πρόκειται για τις δυνάμεις του Μισελ Ντοντοτζά, δημιουργήθηκαν το 2012, είναι κυρίως μουσουλμάνοι. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό όταν σας μιλήσω <clears throat> ειδικότερα για αυτούς τους οποίους στηρίζουμε επί τόπου. Από τους 7.000 που υπήρχαν και ζούσαν σε διάφορα στρατόπεδα, κυρίως κοντά στο Μπάγκι, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν περίπου 1.500 άτομα που σήμερα είναι ενεργά κινούνται προς βοράς, κάποιοι άλλοι αντίθετα. Έχουμε την εντύπωση ότι θα ήθελαν να ενταχθούν σε μια πολιτική διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει. Όταν ε, αναφερόμαστε τώρα στους αντιμπαλακά, Αντίθετα με τους Σελέκα πρόκειται για πολύ βίαιους, ετερόκλητα θα έλεγα, ε, ετερόκλητη σύσταση αυτών των ομάδων. Πρόκειται για μικροεγκληματίες, μικροαπατεώνες, οι οποίοι ουσιαστικά με πλήρη έλλειψη οργάνωσης δημιουργούν αυτές τις ομάδες. Είναι πρώην οπαδοί του Μποζιζέ, υπακούν σε έναν πρώην υπουργό δηλαδή, χωρίς οργάνωση όμως επαναλαμβάνω και σε κάθε περίπτωση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σίγουρα ε, δεν τους δίνει μεγάλη νομιμότητα, είναι παρόλα αυτά επικίνδυνο. Υπάρχουν και πολλές άλλες ομάδες, όπως ξέρετε η πόλη του Μπάγκη σήμερα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει κεντρική διοίκηση, κρατικές ε, ε, αρχές και πολλές φορές οι γαλλικές δυνάμεις βλέπουν σήμερα κάποιες ομάδες να παρουσιάζονται και να επικαλούνται κάποια κινήματα. Υπάρχει μεγάλη, αν θέλετε, βία και εκδίκηση κατά τον ε, Σελεκά από μέρους όλων αυτών των ομάδων. Εκδίκηση, βία και λαιλασία είναι η καθημερινή κατάσταση που επικρατεί ε, σε αυτή την περιοχή. Ο κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει και αυτό που πραγματικά βλέπουμε είναι ότι οι δυνάμεις της γαλλικής επιχείρησης Μίσκα προσπαθούν να ελέγξουν όχι μόνο την πόλη του Μπάνκι αλλά και όλη την ε, επικράτεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Η προστασία των ε, πολιτών η επαναφορά σε μια δημόσια τάξη και η σταθερότητα. Αυτή είναι η εντολή των γαλλικών δυνάμεων. Ενίσχυση δηλαδή της επιχείρησης Μίσκα. Γι' αυτό και σας μιλώ πολύ συχνά για μικτές περιπολίες, για μικτές ομάδες και όσο φυσικά αυξάνεται ο αριθμός των δυνάμεων της Μίσκα, τόσο δυσκολεύει κατά κάποιο τρόπο και ο ρόλος των Γάλλων που βρίσκονται επιτόπου. Σήμερα η επιχείρηση Μίσκα που προέρχεται από μια παλαιότερη επιχείρηση την Μίσκο Παξ 40 άτομα ήταν παλαιότερα και σήμερα οι αξιωματικοί που βρίσκονται εκεί έχουν μείνει 14 με 16 μήνες επιτόπου. 4.700 άντρες, των οποίων ο ρόλος, όπως είδατε από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι η διασφάλιση στην πόλη του Μπάγκη και γύρω από την πόλη. 3.500 ή 3.700 άτομα βρίσκονται στην πόλη του Μπάγκη, οι υπόλοιποι 1.200-1.500 στις ε, υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της ε, Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Τι μπορούμε να πούμε έτσι με έναν απλοϊκό τρόπο. Δεν υπάρχει γενικό επιτελείο, δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει διεύθυνση επιχειρήσεων, δεν υπάρχει διοικητική μέρημνα με την έννοια ότι δεν υπάρχει και αρκετός εξοπλισμός, δεν υπάρχει οργάνωση η κατάσταση, ναι, μεν βελτιώνεται, αυξάνονται οι αριθμοί, με πολύ κακή όμως διαχείριση. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, εξοπλισμός. Δεν μπορούν να κινηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ούτε μέσα στην πόλη, ούτε εκτός της πόλης του Μπάγκη. Επιχείρηση Σάγκαρης, 1600 άτομα που φυσικά εργάζεται υποστηρίζοντας την επιχείρηση Μίσκα. Κυρίως τις πρώτες εβδομάδες σκοπός της ήταν ο έλεγχος της πόλης, από κοινού βεβαίως με την Μίσκα, όχι μόνο στο σύνολο βεβαίως των ε, συνοικιών της πόλης του Μπάγκη. Ελέγχουμε περίπου τα τρία τέταρτα της πόλης. Υπάρχουν ακόμα πολλές συνοικίες οι οποίες δεν ελέγχονται και φυσικά η Μπινούκα που είναι το γραφείο επιχειρήσεων των ε, Ηνωμένων Εθνών για την Κεντροαφρικανική Ένωση. Περίπου 250 άτομα, κυρίως από το Μαρόκο, αποτελούν την ομάδα αυτή Μπινούκα, εντοπίζοντας τη δράση τους τις περισσότερες φορές ε, στα στρατόπεδα που βρίσκονται οι άνδρες της Μπινούκα. Η προβολή των δυνάμεων της Μίσκα. Βλέπετε στην διαφάνεια αυτή το χάρτη και πώς καλύπτουν οι δυνάμεις. 3.500 άτομα στην πόλη του Μπάνκι και 1.500 περίπου που καλύπτουν την υπόλοιπη επικράτεια της χώρας. Δεν μπαίνω τώρα στα, στις λεπτομέρειες της δομής. Ήθελα να σας πω ότι η Μίσκα όσον αφορά τους άντρες που την αποτελούν, πρόκειται για τάγματα τα οποία είναι εξαιρετικά επαγγελματικά. Πρόκειται για επαγγελματίες, επαγγελματικές ενόπλες δυνάμεις. με πολύ ελλειπή εξοπλισμό, όπως σας είπα. Μέχρι τώρα οι εντολές δίνονται μέσω κινητών τηλεφώνων. Ελπίζουμε οι Αμερικανοί να ανταποκριθούν στο αίτημά μας και να καλύψουν τις επικοινωνίες. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η προβολή αυτών των ενόπλων δυνάμεων γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Επανέρχομαι στο προηγούμενο χάρτη για να δείτε ότι ο ομφάλιος λόρος ουσιαστικά είναι ένας δρόμος ο οποίος ξεκινάει από την πόλη του Μπάγκη και κατευθύνεται προς Βοράν. Από εκεί περνάνε όλες οι δυνάμεις. Πώς Μπορεί κανείς λοιπόν να οργανώσει μια επιχείρηση με αυτές τις δυνατότητες. Θα φτάσουμε μέχρι τους 6.000 άνδρες, δηλαδή ένα γενικό επιτελείο το οποίο θα πρέπει να έχει δομή. Επαναλαμβάνω, χρειάζονται ακόμα οχήματα και επικοινωνίες και αυτό προτίθεται να το καλύψουν οι Αμερικανοί. Φυσικά θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να μπορούν να καλύψουν και τις περιοχές εκτός της πόλης του Μπάγκη, καθότι σήμερα η υπόλοιπη χώρα συνεχίζει να είναι ανεξέλεγκτη όσον αφορά την ασφάλεια. Η παρουσία και ο έλεγχος φυσικά και θα γίνει με την αναδιάρθρωση κάποιων ε, ταγμάτων που θα πρέπει να καλύψουν τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό έχει ήδη ε, σχεδιαστεί. Στην χώρα επικρατεί ακόμα ατιμορρησία, συνεχίζει να υπάρχει εγκληματικότητα, κάτι που σαφώς θα μπορέσει να ρυθμίσει μόνο η ύπαρξη αστυνομικών δυνάμεων. Επαναλαμβάνω ότι η επιχείρηση Μίσκα σήμερα περιλαμβάνει μια συνιστόσα αστυνομικών μόνο 630 άντρες. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί αυτή η αστυνομική δύναμη, η οποία βεβαίως επαναλαμβάνω είναι επαγγελματίες και πολύ υψηλού επίπεδου. Πρόβλημα λοιπόν οργάνωσης, υποστήριξης, διοικητικής ε, μέρημνας. Περιμένουμε αυτά που έχουν υποσχεθεί οι Αμερικανοί και φυσικά θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη και η διοικητική μέρημνα μέσω αυτού του άξονα που ξεκινάει από το Καμερούν. Πρέπει να σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 300 οχήματα τα οποία δεν μπορούν να προχωρήσουν, είναι μπλοκαρισμένα καθότι συνεχίζουν οι επιθέσεις, οι δολοφονίες και η λαιλασία στην, στο δρόμο αυτό. Επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο άξονας είναι καθοριστικός για την επιτυχία μιας τέτοιας επιχείρησης, η οποία σημειωτέων έχει ε, στην πρώτη της φάση διήρκησε μόνο τρεις ημέρες. Τώρα, η Ρουάντα έχει στείλει πάνω από 400 άνδρες, θα στείλει άλλους 400 επαγγελματίες. Εξάλλου το πρώτο τμήμα των ενόπλων δυνάμεων της Ρουάντα πέρασε από αυτόν τον άξονα, αυτό το δρόμο. Κατόπιν η εκεί δημοκρατία του Κονγκό, που όπως ξέρετε υποσχέθηκε ότι θα στείλει δυνάμεις οι οποίε δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται στο ίδιο χώρο με τι δυνάμει από την Ρουάντα. Όπω είδατε, υπήρχαν και οι ένοπλες δυνάμεις από το Τσάντ με μεγάλα προβλήματα με τους πρώην Σελέκα. Αυτά βεβαίως σήμερα έχουν ρυθμιστεί. Εδώ θα σας μιλήσω για τις γαλλικές δυνάμεις. 1.600 άνδρες. Βλέπετε και το χάρτη της Γαλλίας για να καταλάβετε πόσο μικρή είναι η Γαλλία σε σχέση με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. 1.600 άνδρες, εκ των οποίων οι περισσότεροι βρίσκονται στη πόλη του Μπάγκη, Εκεί βρίσκεται και το μεγαλύτερο πλήθο, ε, τμήμα του πληθυσμού, καθώς και στην πόλη Μποσανγκόα. Σήμερα έχουμε ενισχύσει τις ε, θέσεις μας και μπορούμε να προβάλλουμε κάποιες δυνάμεις όσον αφορά τον έλεγχο του μεγάλου δρόμου που σας έδειξα, του άξονα αυτού από τον οποίο περνάνε όλες οι δυνάμεις. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές. Θα σας μιλήσω για την πόλη Μπριά που βρίσκεται ανατολικά, την περιοχή Σίμουτ, βόρεια του Μπάνγκη αλλά και την πόλη του Μπουάρ με πολλά προβλήματα βίας στις περιοχές αυτές. Να σας υπενθυμίσω επίσης, για να καταλάβετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί και την κατάσταση των γαλλικών δυνάμεων, ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν έχουν καλύψει το υπόλοιπο, την υπόλοιπη επικράτεια. Εμείς είχαμε αναλύσει την κατάσταση που φυσικά δεν ήταν καινούργια, απλώς είχε επιδεινωθεί χάρη σε κάποιες προληπτικές ε, δράσεις και επιχειρήσεις. Είχαμε καταλάβει ότι αν έπρεπε να υπάρξει προβολή γαλλικών δυνάμεων, το κεντρικό σημείο θα έπρεπε να είναι το αεροδρόμιο. Έπρεπε να γίνει μια σχετική βελτίωση της κατάστασης της ε, πίστας. Φτάσαμε στις 5 Δεκεμβρίου και υπήρξε μία σχετική προετοιμασία επιτόπου. Οι γαλλικές δυνάμεις έφτασαν διαθαλάσσεις ε, στο Καμερούν και στο Γκαμπόν. Από το Δεκέμβριο ήδη ξεκίνησε η πρώτη επιχείρηση. Φυσικά εδώ χρειάζεται κινητικότητα, χρειάζονται προτεραιότητες. Όλα αυτά αντιμετωπίζοντας πολύ σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά την επιχείρηση Μίσκα, την οποία καλούμεθα να υποστηρίξουμε, με προβλήματα σχεδιασμού, με προβλήματα διοίκησης, με προβλήματα οργάνωσης. Σήμερα βέβαια όλα έχουν ε, ρυθμιστεί και εξομαλυνθεί. Περίπου 10 Γάλλοι αξιωματικοί επιτόπου στήριξαν την επιχείρηση Μίσκα βελτιώνοντας τις δυνατότητες διοίκησης των επιχειρήσεων. Εδώ βλέπετε τις κινήσεις των γαλλικών δυνάμεων από το Καμερούν και από τον Καμπόν προς την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες της επιχείρησης Σάγκαρης. Αυτά που σας είπα νομίζω αρκούν υποστήριξη του Γενικού Επιτελείου, πληροφορίες, αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις θα επανέλθω σε αυτήν την διαφάνεια. Για μας η κατάσταση σήμερα είναι σχετικά σταθεροποιημένη. Βλέπουμε δυνάμεις να φεύγουν προς βοράς με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι διάφορες ε, δραστηριότητες των πρώην ΣΕΛΕΚΑ που σήμερα επαναλαμβάνω ελέγχονται από τις γαλλικές δυνάμεις και από την επιχείρηση ΜΙΣΚΑ. Είναι επικίνδυνο βεβαίως το ότι υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση στην περιοχή Μπριά. Γι' αυτό ακριβώς και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι γαλλικές δυνάμεις ή οι δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που ελέγχουν την ε, επιχείρηση Μίσκα θα μπορέσουν να επεκταθούν και να καλύψουν τις υπόλοιπες περιοχές, τις υπόλοιπες πόλεις και να ελέγξουν και τις δραστηριότητες των πρώην Σελέκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ στρατηγέ. οι αρχές της επέμβασης έγιναν δεκτές ε, τη Δευτέρα στο Συμβούλιο ε, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη φάση του σχεδιασμού. Να ακούσουμε λοιπόν τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω συντομία τα βασικά στοιχεία της απόφασης αυτής ε, του Συμβουλίου, πατώντας στο αίτημα του Πρόεδρου. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία και θα σας πω που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την προπαρασκευαστική αυτής της επέμβασης και ποια είναι τα επόμενα στάδια. Τι αποφάσισε λοιπόν το Συμβούλιο. Έλαβε την πολιτική απόφαση να γίνει τη Δευτέρα συγκεκριμένα, να γίνει αυτή η επιχείρηση με βασικό στόχο να εξασφαλιστεί η προστασία των αμάχων και να συνεισφέρουμε και εμείς ε, σε όσα προβλέπονται από το ψήφισμα 21-27 της για να αποφύγουμε την επιθύνωση της κατάστασης και για να στηρίξουμε την πολιτική διαδικασία η οποία φαίνεται να διαγράφεται. Δύο είναι τα βασικά συμφέροντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα το θέμα της προστασίας των αμάχων ε, και για να μην ε, υπάρχει κίνδυνος γενοκτονίας. Πολλοί εκπρόσωποι των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες κάνουν λόγο για μια κατάσταση ε, προ-γενοκτονίας. Και ένα δεύτερο διακύβευμα να μην υπάρξει μετάδοση στην, επόμενη, στην υπόλοιπη περιοχή, γιατί η περιοχή αυτή γενικά παραμένει ευάλωτη και η κατάσταση είναι ρευστή. Τι αποφάσισε το Συμβούλιο, τι προτείνεται και σε τι θα συνίσταται αυτή η ε, επέμβαση. Πρώτα απ' όλα, στήριξη της ΜΙΣΚΑ και της γαλλικής επιχείρησης ε, με μια παρουσία ασφαλείας στον Παγκουή ε, για να συμβάλλουμε και εμείς στη σταθεροποίηση της χώρας και στην προστασία των αμάχων. Πρώτη πτυχή αυτή με βάση ε, τον τρόπο δράσης που περιβά, γράφηκε. Θα προσπαθήσουμε και αυτή τη φορά να έχουμε μια παρουσία ασφαλείας στον Παγκού. Η δεύτερη πτυχή της ε, επιχείρησης, της αποστολής αυτής ε, που θα διευκρινιστεί σε συνεργασία και με την Αφρικανική Ένωση είναι και στην περίπτωση αυτή να στηρίξουμε την ΜΙΣΚΑ ώστε η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης να μπορέσει το συντομότερο δυνατόν να φέρει αποτελέσματα και να αναλάβει την αποστολή της σταθεροποίησης και της ασφάλειας. Συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο για αυτή την επιχείρηση ε, η διάρκεια της αποστολής να είναι έξι μήνες από τη στιγμή που θα αναπτύξει επιχείρηση επιχειρησιακή δυνατότητα. Και τελευταία σημαντική παράμετρος, το Συμβούλιο αποφάσισε κυρίως για λόγους ανθρωπιστικούς και προστασίας των αμάχων η αποστολή να εστιάσει στην περιοχή του Μπάνγκουι. Εκεί δηλαδή που είναι οι περισσότεροι εκτοπιστέντες, έχουμε το ζήτημα του αεροδρομίου και του καταφυλισμού των προσφύγων με πάρα πολλέ χιλιάδες ανθρώπους, είναι πρόβλημα. Ε, υπάρχουν λοιπόν παράμετροι, το αεροδρόμιο κτλ. που μας κάνουν να θεωρούμε ότι καλό είναι να εστιάσουμε σε αυτή την περιοχή του Μπαγκούι. Αυτή η επέμβαση παρασκευάζεται σε στενή συνεργασία και συντονισμό με όλου του εταίρου μα από τη διεθνή κοινότητα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. ξεκινώντα από την Αφρικανική Ένωση, είχαμε και άτυπε επαφέ, έγιναν κάποια διαβήματα και από την προσωπία μα στην αντί. Υπάρχει τώρα ε, και μια ε, αντιπροσωπή ε, αποστολή της ΕΙΕΔΕ στην Αντίς και συζητάει το θέμα αυτό. Επίσης, στον Παγκού είχαμε επαφές και με τον στρατηγό Γκαρσία και με τον στρατηγό Μοκόκο, εκπρόσωπο της Αφρικανικής Ένωσης. Και ε, οι δύο στρατηγοί, Γκαρσία και Μοκόκο, δήλωσαν ότι στηρίζουν ε, πλήρως αυτή την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βέβαια, είχαμε πολύ στενή συνεργασία και με τα Ηνωμένα Έθνη, ο Γενικός Γραμματέας και το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκαν με επιστολή της κυρίας Άστον από τη στιγμή μάλιστα που ελήφθη η απόφαση του Συμβουλίου είχε ενημερωθεί ε, ο ΙΕ Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μετά τον Νοέμβριο για τις υπηρεσίες ε, διατήρησης της ειρήνης ε, που έχουμε. Υπάρχει λοιπόν απόλυτη στήριξη αυτής της ε, αποστολής. Χθες συνεδρίασε του Συμβουλίο Ασφαλή, αν δεν ο ειδικό εκπρόσωπος του ΓΑΜΑΓΑΜΑ των ΟΕΕ Εθνών για το ζήτημα των παιδιών ε, σε εμπόλεμες περιοχές και το Ειδικό ε, Συμβούλιο για την πρόληψη της γενοκτονίας, ο ειδικό εκπρόσωπος του Γενικού για τη σεξουαλική κακοποίηση. Όλοι στήριξαν ε, την ιδέα της επιχείρησης αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτος εταίρος βέβαια η ίδια η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ενημερώθηκε βέβαια τηρείται ενημερή όλη αυτή τη διαδικασία και επισήμω με επιστολή τη κυρία Άστον, όταν ελήφθη από το Συμβουλίο, ενημερώθηκε και την και Δημοκρατία όλε τι επαφέ που είχαμε είτε έχουμε την αποστολή στον Πάγκο, όπως σας είπα, ε, γίνονται δεκτές θετικά από την πλευρά της Κεντρικής ε, Αφρικής. Και έχει στέλνει και επιστολή στην στον ΟΗΕ από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που επίσης δηλώνουν την υποστήριξή τους οι αρχές σε αυτή την αποστολή. Σε ό,τι αφορά τώρα το συντονισμό της ε, ευρωπαϊκής οικογένειας και με το ΕΚΟ είχαμε ε, επαφές ήδη ευθύς εξ αρχής. Από την αρχή έχουμε συνεργαστεί τα έγγραφά μας ε, τα ανταλλάσσουμε για να μην σας πω ότι ε, τα καταρτίζουμε και οι δύο μαζί. Και πρέπει να σας εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για αυτή την τόσο καλή διαδικασία συντονισμού. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ένα έγγραφο και ένα ε, έγγραφο σχεδιασμού που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας και βέβαια υπάρχει και η απαραίτητη αυτονομία για να μπορέσει να ασκηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η επιχείρηση. Αυτά σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους. Πού βρισκόμαστε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η απόφαση της Δευτέρας είναι μια πολιτική απόφαση για δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ετοιμάσει μια αποστολή και αυτό θα γίνει με, την, με τον ορισμό μιας έννοιας διαχείρισης κρίσεως, ενός κόνσεπτ διαχείρισης κρίσεως. Έχουμε τώρα δύο γραμμές δράσης, σήμερα μην πω τρεις, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να τις επεξεργαζόμαστε. Πρώτον, πρέπει να ορίσουμε το νομικό πλαίσιο του στο οποίο θα διεξαχθεί αυτή η επιχείρηση. Και θα ξεκινήσουμε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τις επόμενες ημέρες το Συμβουλίο Ασφαλείας θα συνεδριάσει για να αποφασίσει την επέκταση της ε, εντολής της ε, Μπιμούκα θα είμαστε σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη και η κυρία Άστον, βέβαια έστειλε επιστολές στον πρόεδρο της Συμβουλίου Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα, για να τους μεταφέρει την απόφαση του Συμβουλίου. Δεύτερη πτυχή του νομικού πλαισίου, απόφαση του Συμβουλίου, επίσημη απόφαση που είναι η νομική βάση στο εσωτερικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την επέμβαση. Ξεκίνησαν οι σχετικές εργασίες και περιμένουμε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μηνός. Τρίτο στοιχείο σε αυτό το νομικό πλαίσιο, συμφωνία ε, για το καθεστώς των δυνάμεων με τις κεντροαφρικανικές αρχές είμαστε σε επαφή. Μας είπαν δεν έχουν δυσκολία, μπορούν να μας δώσουν ε, τα απαραίτητα προνομιά και ασυλίες. Για την ιστορία να σας πω ότι ήδη είχαμε με την κεντροαφρικανική δημοκρατία μια τέτοια συμφωνία όταν επιχειρήσαμε στο Τσάντα. Είναι γνωστό δηλαδή το πεδίο και το έχουμε χαρτογραφήσει και οριοθετήσει. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή δραστηριότητας. Δεύτερη, σχεδιασμός, επιχειρησιακός σχεδιασμός, δηλαδή η πολιτική αυτή πρόθεση που εξέφρασε στο Συμβούλιο πρέπει να μεταφραστεί σε επιχειρησιακό σχεδιασμό που θα ε, περιγράφει συγκεκριμένα το πώς θα ε, πραγματοποιηθεί αυτή η επιχείρηση. Από τις Βρυξέλλες λοιπόν θα περάσουμε πλέον ε, στη διοίκηση. Θα ορίσει βέβαια η, θα ορίσουν οι Βρυξέλλες ποια θα είναι τα μέλη. Και έτσι θα φτάσουμε σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα πρέπει να εγκρίνει το Συμβούλιο. Ελπίζουμε αυτό να γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Και εν συνεχεία θα έχουμε την παραγωγή δυνάμεων, δηλαδή θα εντοπιστούν οι χώρες που μπορούν να συνεισφέρουν και θέλουν να φέρουν στρατεύματα, να συνεισφέρουν τα στρατεύματά τους. Βέβαια θα πρέπει και τη διοίκηση, την αλυσίδα διοίκηση να την ε, ορίσουμε. Προχωράμε καλά και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την αλυσίδα της δίκησης θα ξέρουμε σύντομα ποιοι θα είναι αυτοί. Για τους ε, συνεισφέροντες, επόμενες ε, ημέρες θα οργανωθεί ε, μία συνέλευση για να οριστούν, να εντοπιστούν οι χώρες που θέλουν να συνεισφέρουν. Υπάρχουν και ανεπίσημες επαφές ήδη, για να έχουμε την κρίσιμη μάζα των χωρών που θα παρτίσουν αυτή την επιχείρηση. Τρίτον, ενημέρωση των εταίρων. Ενημερώσαμε βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τους βασικούς μας εταίρους, Αφρικανική Ένωση, ΗΠΑ ε, και οι Έθνη που έλαβαν επιστολή. Επίσης, με βάση τη Συμφωνία Συντονισμού, στείλαμε και στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ μια επιστολή να τον ενημερώσουμε για την απόφαση του Συμβουλίου. Δημερός, επίσης, ενημερώσαμε ορισμένε χώρες οι οποίες συνήθως συμμετέχουν στις επιχειρήσεις μας, τρίτες χώρες, Καναδάς, Νορβηγία, Τουρκία και συνεχίζουμε ε, ενημερώνοντας και τις χώρες της περιοχής. Με τους πρέσβεις θα συναντηθούμε για να τους ενημερώσουμε και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης. Στόχος είναι οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν κατανοητές και να εκφραστούν ε, σωστά για τα battle groups τώρα, αυτούς τους σχηματισμούς μάχης. Τρεις, σε τρει χρόνους θα απαντήσω. Πρώτον, μπορούσαμε να τα είχαμε χρησιμοποιήσει τα battle groups για αυτή την επιχείρηση. Από τεχνική πλευρά, αυτή η έννοια δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην επιχείρηση όπως εμείς την σχεδιάζουμε. Τα battle groups είναι για 120 ημέρε. Εμείς θέλουμε να είναι λίγο ε, πιο μεγάλος ο χρονικός ορίζοντας. Επίσης, μπαίνουν στο θέτρο επιχειρήσεων αυτές οι ομάδες... ενώ εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Η ταχύτητα όμως ε, ε, και επιθέλαμε να είμαστε και ευέλικτοι, μας ε, έκανε να ε, μην προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήταν δυνατόν όμως να την είχαμε χρησιμοποιήσει, αν και δεν είναι ακριβώς αυτό που αντιστοιχεί. Τώρα, η κοινή πολιτική άμεση και ασφάλεια είναι διακυβερνητική πολιτική, όπω είναι προφανή, και τα κράτη-μέλη είναι προσιλωμένα στο να παραμείνει έτσι η κατάσταση. Προτού λοιπόν χρησιμοποιήσουμε στρατεύματα από μια χώρα, καλό είναι ε, από πολιτικής πλευράς να ρωτήσουμε τη χώρα αν θέλει κάτι τέτοιο. Είχαμε λοιπόν επαφές και τον Νοέμβριο με τις χώρες που συνεισέφεραν ε, στους σχηματισμούς μάχης και είχαν ενημερωθεί τον Νοέμβριο και επίσης την 1η Ιανουαρίου. Λάβαμε λοιπόν, ε, είχαμε τις επαφές, χώρες αυτές μας είπαν ότι θα προτιμούσαν να συμφέρει στο πλαίσιο ε, μιας επίσημης δικασίας συγκρότησης δυνάμεων Άρα δεν μπορούσαμε να προτείνουμε κάτι το οποίο δεν θα ήταν σύμφωνο με την άποψη των κρατών μελών, ένα battle group δηλαδή. Τώρα αν είναι ικανοποιητική η απόφαση, 100%. Ε, Πρέπει να σας πω ότι Φυσικά και δεν είναι 100%, αλλά μια απόφαση του Συμβουλίου το Δεκέμβριο ήταν ακριβώ να εργαστούμε ώστε αυτή την έννοια του Battle Group να την κάνουμε πιο ευέλικτη, να μπορεί να τροποποιείται, να είναι πιο εύπλαστη, αν μπορώ να το πω έτσι και να μπορεί μια χώρα όταν δεν θέλει να συνεισφέρει να αντικαθιστεί από μια άλλη. Στις 20 Δεκεμβρίου λοιπόν το κόνσεπτ αυτό ε, ξεκινήσαμε να το εξετάζουμε, είμαστε 23 Ιανουαρίου, δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα, συνεχίζονται οι συζητήσεις, ξεκίνησε όμως η διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα δούμε τι καρπούς θα φέρει, ας περιμένουμε. Πώς το παρόν αυτά είχα να πω, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για να συμπληρώσουμε αυτό το επιχειρησιακό τοπίο έπρεπε να δούμε και την πολιτική σκοπιά όλου αυτού του πλαισίου. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος, εφόσον είχατε μια πολύ ε, συνοπτική παρουσίαση, ε, πολύ σφαιρική για την ε, συνολική κατάσταση. Είναι πολύ σημαντική η κατάσταση. Είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αυτή, διότι η εκλογή της Προέδρου για την προσωρινή κυβέρνηση δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσει μια πολιτική διαδικασία και να βρεθεί ενδεχομένω διέξοδο από, την, ε, από τις εχθροπραξίες και την σύγκρουση που θα μπορούσε να ξεφύγει τελείω από κάθε έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνεί στρατιωτικέ δυνάμει βεβαίω που είναι παρούσα στη χώρα θα πρέπει να παράσχουν ασφάλεια προκειμένου αυτή η πολιτική πορεία να ξεκινήσει απρόσκοπτα. Αυτό προσπαθούν η Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα και η Αφροκανική Ένωση με την ε, ε, δύναμη της την Μίσκα προσπαθούν να κάνουν. Ακούσατε πώς έχει κατάσταση εσωτερικής ασφάλειας, η οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ακόμη και από τότε που είχαμε 3.500 ε, άνδρες της Μίσκα στο Μπανγκή Ακόμη και από την εκλογή της κυρίας Κάθριν Σαμπαπάντζα και μετά συνέχισαν να υπάρχουν ε, εχθροπραξίες και θάνατοι στον Μπάνγκη και βεβαίως και στην υπόλοιπη χώρα. Η, ε, ε η Σελέκα, η, αντι, η Αντιμπαλάκα επίσης ε, συνεχίζουν να είναι εχθρικοί μεταξύ τους και υπάρχουν πολλοί εκτοπισμένοι. Οι συνθήκες είναι δύσκολες για να υπάρξει μια πρόσκοπτη και ομαλή πολιτική διαδικασία, κυρίως γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες, συστηματισμοί ή και ηγέτες. Χρειάζεται λοιπόν σχηματισμοί η χώρα αυτή. Το πρόβλημα ε, είναι σύνθετο όμως, διότι όπως είπε και η Επίτροπος Γεωργίευα, η κοινωνική κατάσταση έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη. Ο κοινωνικός ιστός αρχίζει να διαρριγνύεται. Οι διαφορές μεταξύ των κοινοτήτων δεν είναι μόνο οι διαφορές μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, είναι μεταξύ αστών ε, εντός εισαγωγικών και γεωργών, είναι μεταξύ βορρά και νότου. Ε, υπάρχει λοιπόν μια διαρκή στάση αντιπαράθεσης η, πολι... η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, αλλά μόλις αυτή ε, ε, εξασφαλιστεί, τότε θα πρέπει να υπάρξουν ε, περισσότερες πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες. πρέπει να υπάρξει δράση. Η Πολιτική Επιτροπή σήμερα μίλησε στους θρησκευτικού ηγέτες της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, χριστιανούς και μουσουλμάνους που βρίσκονταν εδώ, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλέστερο, ειρηνικότερο περιβάλλον. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι επίσης και πώς θα δεσμευτεί η διεθνής κοινότητα. Η σύνοδος του ΕΚΑΣ που οδήγησε στην απόσυρση του προηγούμενου Προέδρου και της κυβέρνησης έδωσε την ε, δυνατότητα για όλη αυτή τη διαδικασία. Οι γειτονικέ χώρες, η διεθνή κοινότητα και η Αντροαφρικανική Δημοκρατία προσπαθούν να έχουν μια ενιαία συντονισμένη προσπάθεια για να ευοδοθεί αυτή η πολιτική πορεία. Πράγμα που θα συνεχιστεί και στη Σύνοδο της Αφρικανικής ε, Ένωσης την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό όμως το κατά πόσο θα δεσμευτεί η ΕΚΑΣ, γιατί οι γειτονικές χώρες όλες πλήττονται από την κρίση της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας, όλες ανησυχούν για τις περιπτώσεις να υπάρξουν συνέπειες και στις ίδιες με πρόσφυγες, με εχθροπραξίες και στα δικά τους ε, εδάφη και πραγματικά έχουν άμεσο συμφέρον στο να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ειρηνική πολιτική διαδικασία με κυβερνητικές δομές σταθερές στη χώρα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε μαζί με τους ανθρώπους της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, της Αφρικανικής Μέλλον ε, για να βρεθεί μια διέξοδο όπως έχουμε κάνει και σε άλλες ε, περιστάσεις. Η πολιτική μας λοιπόν ε, παρέμβαση έγκυται στο να στηρίξουμε την κυβέρνηση και την ειρηνική πολιτική διαδικασία σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τον στρατηγό ΚΑΙ, ο οποίος είναι επίσημος εκπρόσωπός μας εκεί με τα στρατεύματά του. Στο βαθμό στον οποίο μπορούμε να δαπανίσουμε κονδύλια της ανάπτυξης προκειμένου να έχουμε αναδόμηση των κυβερνητικών δομών, να αρχίσουν οι άνθρωποι να δουλεύουν και πάλι, ε, να παίρνουν και το μισθό τους, να λειτουργούν τα τελωνία και ούτω καθεξής, είναι ήδη σημαντικό. Η αντιπροσωπεία μα που καθ' όλη τη διάρκεια τη κρίση στον Πανγκή έχει παρακολουθήσει τι εξελίξει, είναι σε στενέ επαφέ με, ε, με τι αρχέ για να δουν τι μπορεί να γίνει. Εργάζονται σε συνεργασία με την ΔΕΦΚΟ και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από τον προπολογισμό για την ανάπτυξη, από το εργαλείο για τη σταθεροποίηση, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τι εκεί ανάγκε αλλά πρέπει και η κεντροαφρικανική δημοκρατία να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε το κράτος να μπορέσει να ε, πατήσει στα πόδια του και να αρχίσει να περπατά. αυτά είχα να πω και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις διευκρινήσεις. Πολλοί βουλευτές ε, θέλησαν και ζήτησαν το λόγο για αυτή τη συζήτηση. Η κυρία Γκόμες πρώτα. Κάποιες ερωτήσεις προς εσάς ε, ταξιερχέ και εσάς κύριε Βαστκούτ. Πιστεύετε ότι ο κίνδυνος γενοκτονίας έχει αναχαιτιστεί, έχει αντιμετωπιστεί κάπως λόγω των εξελίξεων που αναφέρατε. Πιστεύετε ότι αποφύγαμε τον κίνδυνο της ε, της της μετάδοσης αυτής της ε, σύγκρουσης και εκτός των συνόρων. Ε... Μπορεί δηλαδή να ξεφύγει από τα σύνορα της χώρας η ένταση και για την ε, επιχείρησή μας. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί. Θα παρακολουθήσουμε τον επιθανάτιο ρόγχο της ανάγκης αυτής να υπάρξει άμεση παρέμβαση, επέμβαση μάλλον, ενώ τα κάτι μέλη θα ολιγορούν διότι το πρόβλημα δεν είναι η διοργάνωση μας σε επίπεδο Βρυξελών, αλλά σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό παίρνει πολύ χρόνο. Και εν τέλει, να σα ρωτήσω, δεν ξέρω αν θα μου απαντήσετε εσείς εσεί ή εσείς Βέσκο, η κυριε λενουαρ διάσταση, τα διαφορετικά δόγματα. Το συζητάμε πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι ε, αντικείμενο πολιτικών σκοπιμοτήτων τη πράλης. Εδώ BBC έναν ε, κύριο ο οποίο έλεγε ότι είναι χριστιανό και εξηγούσε πώ έφαγε την καρδιά και τα άλλα όργανα ενός μουσουλμάνου γιατί του είχε σκοτώσει την οικογένεια εκείνος. Ε, τώρα τι σημασία έχει ένα χριστιανοί μουσουλμάνοι, έτσι. Δεν πολύ πιστεύω σε αυτά. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν δύο λόγια γι' αυτό, για τις θρησκευτικέ διαφορές. Ευχαριστούμε, Άννα. Ο κύριος Φανόρντον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε δεδομένου του χαρακτήρα και της κλίμακας και μάλλον και του κατεπήγοντος χαρακτήρα της ανάγκης επέμβασης θα ήταν απλούστερο οι γαλλικές δυνάμεις να αναλάβουν τη γενική, το γενικό συντονισμό θα αναλάβει ο, ε, να τον αναλάβουν στο Σαν παρά όπως γινόταν ως τώρα να συντονιστεί όλα αυτά από τη Γιουνίσα και χωρίς να υπάρχουν καλοπιστικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να είναι περιττές. Βέβαια μπορεί να υπάρξουν και στρατεύματα που θα πάρουν μέρος και δεν θα είναι Γάλλοι, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το τι εννοούμε για την επιχείρηση. Ε, ο στόχος είναι να υπάρξει επικράτηση ασφαλείας στο Μπανγκί. Τι θα γίνει στην υπόλοιπη ποια δύναμη θα αναλάβει την ε, σταθεροποίηση στον Παγκία αυτή που είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο θα είναι μόνο αμυντικός ο ρόλος της ή θα προσπαθήσει και σε άλλα μέρη της χώρας να αναλάβει δράση. Και επίσης με ενδιαφέρει ποια είναι η προοπτική μας για το μέλλον. Λέτε ότι μιλάμε για μια εξάμεινη επιχείρηση. Μετά από έξι μήνες ποια ε, θέτεται ότι μπορεί να είναι η κατάσταση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Θα τον δώσετε, θα δώσετε τη σκητάλη στην Αφρικανική Ένωση μετά από έξι μήνες. Ευχαριστούμε κυρία Λέζινγκ. Ε, ε, Ευχαριστώ η συνάδελφος από την Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, δεν θυμάμαι το όνομά της, είπε πολύ σωστά ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια που έχουν δοθεί για την επιχείρηση Μίσκα και πολύ λιγότερα έχουν δοθεί για την ανθρωπιστική πτυχή αυτής της επιχείρησης. Ο πρόεδρος των γιατρών Χωρίς Σύνορα έστειλε μία επιστολή πριν τα Χριστούγεννα αναφερόμενος στην επίγουσα ανάγκη να συγκεντρωθούν κονδύλια για την χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής πτυχής. Εδώ δεν καταλαβαίνω, χρηματοδοτούμε με αναπτυξιακά κονδύλια στρατιωτικές επιχειρήσεις, μήπως θα ήταν καλύτερα να πάνε κατευθείαν στην ανθρωπιστική βοήθεια αυτά τα κονδύλια. Βεβαίως οι εκπρόσωποι των δημοκρατικών δυνάμεων θα πρέπει να μπορέσουν να εκφραστούν. Το θέμα είναι βεβαίως ότι πολλές φορές αναρωτιόμαστε οι πολίτες, ο λαός αυτών των ε, χωρών μήπως θα πρέπει να ενημερωθούν ότι χρησιμοποιούμε εδώ για να χρηματοδοτήσουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις αναπτυξιακά κονδύλια και αυτά προέρχονται από τον φορολογούμενο. Είναι δικά τους τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον ε, κύριο Λενουάχ. Γιατί μπορούμε να ακούσουμε όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ και μετά μπορούμε να ακούσουμε και τον κύριο Μπόερ ο οποίος είναι υπεύθυνος από την ΕΚΟ ε, για να μας ενημερώσει για τις ανθρωπικές διαστάσεις του θέματος. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα για να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις και μετά για την, επιχείρηση. Θα χρηματοδοτηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και η επιχείρηση Αθηνά, από την επιχείρηση Αθηνά και όχι από κοινοτικά κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν προβλέψαμε ένα μηχανισμό ανάλογο με το Αθηνά. Επίσης, για το αν θα ήταν απλούστερο απλώς οι Γάλλοι να αναλάβουν αυτή την επιχείρηση μόνον δεν νομίζω ότι θα σας πω κάποιο μυστικό εάν σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πίεσε η Γαλλία για να υπάρξει ευρωπαϊκή επέμβαση. Η ΕΕ δεν ε, θέλει να αμφισβητήσει τις πολιτικές κατευθύνσεις που έδωσε, τους πολιτικούς προσανατολισμούς που έδωσε το Συμβούλιο των ε, Πρωθυπουργών και ιδίως ο Γάλλος Πρόεδρος. Τώρα, για το τι προβλέπουμε, κύριοι βουλευτέ, δεν είναι επιχειρησιακή μα ζώνη το ρόδρομο του Μπαγκή. Η συμφωνία του Συμβουλίου αφορά ε, και έχει ακριβώ τη μνήμα in the Bangui area, στην όλη περιοχή του Μπαγκή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει επιχειρησιακό σχεδιασμός από το επιτελείο που παρόλα αυτά έχει αναλάβει την περιοχή του αεροδρομίου. Και υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, κανόνες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό αφού αναλυθεί προσεκτικά η κατάσταση. Και βεβαίω μετά το σχέδιο αυτό θα πρέπει να το εγκρίνει και το Συμβούλιο και έπειτα για το end state, για το τέλος της αποστολής. Μίλησα για ένα εξάμεινο από τη στιγμή που θα αναπτυχθεί πλήρως η στρατιωτική μας δύναμη. Αυτό είναι επίσης σημαντικό ως παράγον. Έξι μήνες από την πλήρη εκτύπωση. Η εκτίμησή μας είναι ότι έξι μήνες μετά και χάρη στη στήριξη της Μίσκα, προς τη Μίσκα μάλλον από τη Γαλλία, που θα μπορούσε να συμπληρωθεί από τους Αμερικανούς ή και την ευρωπαϊκή επιχειρήση, τότε η ΜΙΣΚΑ θα μπορούσε να αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των πτυχών ασφάλειας που αυτή τη στιγμή θα εξασφαλίσει η ευρωπαϊκή επιχειρήση. Μιλάμε για μια σύνδεση λοιπόν των επιχειρήσεων, bundling, με άλλα κομμάτια επιχειρησιακά, κάτι που δεν μπορέσει να αναλάβει εξ τώρα η ΜΙΣΚΑ. Τελευταία παρατηρήση για τις διάρκειες η διαδικασία σχεδιασμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εκδίπλωση των δυνάμεων θα πρέπει να ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώ επί τόπου. Αν όλα πάνε καλά και ο επιχειρησιακό σχεδιασμό γίνει εγκαίρο και υπάρξει και η σωστή εκδίπλωση, εάν δεν υπάρξουν φοβερά προσκόμματα δηλαδή, νομίζω ότι μετά από λίγε εβδομάδε θα μπορούσαμε να έχουμε τα πρώτα βήματα μια ευρωπαϊκή επιχείρηση στον Πανγκή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, κύριε Ταξίρχε. Δύο σημεία να αναπτύξω την ερώτηση της κυρίας Γκόμες για τις θρησκευτικέ διαφορές. και την ε, διευκόλυνση για την ειρήνη στην Αφρική. Αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι υπάρχει σοβαρό κίνδυνο γενοκτονία Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ πολιτών και είναι πολλές οι συνιστώσεις αυτής της σύγκρουσης. Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ κοινοτήτων, εθνοτικές διαφορές, μεταξύ κάποιων που είναι ουσιαστικά αστεί και μουσουλμάνοι και των γεωργών που βρισκόνται στα νότια και δυτικά της χώρας και είναι κυρίως χριστιανοί αλλά όχι αποκλειστικά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές συνιστώσεις παράμετροι στο πρόβλημα. Ο κίνδυνος των εχθροπραξιών μεταξύ των πολιτών που μπορεί να κλιμακωθεί θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενοκτονία και μέχρι να αποκατασταθεί ασφάλεια τα πάντα μπορεί να συμβούν σε εχθροπαξίες μεταξύ ατόμων, πολιτών, ομάδων, ανοργάνωτων, οργανωμένων, παραστατικών. Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει κατάρρευση των σχέσεων εμπιστοσύνης ως τώρα μεταξύ των κοινοτήτων. Αυτή που υπήρχε ως σήμερα και αυτό κάνει να αναφλέγονται οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, οι προσπάθειες συμφιλίωσης μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων και των εθνοτικών ομάδων είναι η μόνη μας ευκαιρία. Οι εκτοπισμένοι πολλές φορές είναι μεικτοί πληθυσμοί, μεικτές ομάδες ανθρώπων, ακόμη και στους στα στρατοπέδα προσφύγων. Είναι διαφορετική προέλευση οι άνθρωποι που συγκατοικούν, συνυπάρχουν στα ίδια στρατόπεδα και καταφέρουν να συνεπάρξουν σε συνθήκε εμπιστοσύνη. Έπειτα, για τη χρήση τη ε, για την ειρήνη στην Αφρική. Όπως είπε και η Επίτροπος Γεωργίευα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τεράστιες προσπάθειες για να στηρίξει την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι, οι ίδιοι υπεύθυνοι για τα ανθρωπιστικά λένε ότι χρειαζόμαστε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για να προσφερθεί αυτή η βοήθεια. Ιδάλλως δεν μπορούμε να την προσφέρουμε. Χωρίς λοιπόν ασφάλεια, οι ανθρωπιστικές μας προσπάθειες εν μέρη είναι αναποτελεσματικές και αρχίζουν να γίνονται και πιο ασαφείς. Δηλαδή μπορεί να περάξουν χρόνια ε, που θα στέλνουμε χρήματα σε στρατοπέδα προσφύγων, αλλά όταν κάποιο δεν μπορεί να πάει πίσω ασφαλώ στι αιστείε του, δεν μπορεί να ε, καλλιεργήσει τα χωράφια του, να κάνει τη σπορά, τη συγκομιδή και να θρέψει τον εαυτό του. Ε, η ανθρωπιστική λοιπόν βοήθεια σημαίνει ότι για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχουμε και πάλι ειρηνικέ συνθήκε, ε, εύρυθμη λειτουργία του κράτου για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια του. Οι προσπάθειες λοιπόν για την ε, ασφάλεια και για την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα. Ε, τα κονδύλια από το Ταμείο για την Ανάπτυξη και για τη στήριξη της ε, διευκόλυνσης της ειρήνης για την Αφρική είναι πράγματα που πρέπει να συνδυαστούν η ασφάλεια με την ανθρωπιστική βοήθεια. Τα κονδύλια όμω αυτά πρέπει να δαπανηθούν τώρα, τώρα να εκταμιευθούν, διότι οι δαλώς οι άνθρωποι αυτοί θα υποφέρουν ακόμη περισσότερο, η κατάσταση θα συνεχιστεί επάπειρον για μήνε και χρόνια. Είναι θέμα επενδυτικό περισσότερο και πραγματικά αυτό θα το προβάλλω ω επιχείρημα και ενώπιον των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Είναι χρήματα που θα δαπανηθούν σωστά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν σωστά τη δουλειά του και να καλύψουν τι δικέ του πια οικονομικέ ανάγκε. Moi, si je peux rebondir sur le risque de génocide, oui. Ευχαριστώ να απαντήσω και εγώ. Κίνδυνο γενοκτονία. Ναι, δεν έχει εκλείψει. Τι εννοούμε όμω με τον όρο γενοκτονία. Μιλάμε για πολυάριθμε ε, πράξει βία. Αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Επιτόπου οι Γάλλοι στρατιώτες και έχουμε πραγματικά πράξεις βίας απίστευτης αγριότητας για να μην σας πω κανιβαλισμό. Όταν έχουμε να κάνουμε ένα τέτοιο, με μια τέτοια κατάσταση βίας είναι πολύ αριθμή κίνδυνη. Αν δεν τα πάει καλά η πολιτική διαδικασία και αν δεν ελέγξουμε τα έκτροπα των ε, Σελέκα, ε, πρέπει να αποφύγουμε ε, τις ε, αντιπαραθέσεις αντιμπαλάκα σε λέκα και αν δεν τα μαζέψουμε κάπως τα πράγματα θα έχουμε ε, ανάφλεξη και υπάρχει κίνδυνος και υποσυτισμού, λιμοκτονίας. Αν κοπεί, αν υπάρχει αυτή η... αυτός ο αποκλεισμός, αν κοπεί αυτός ο ομφάλιος λόρος θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα ιατρικό. Τώρα, η σχέση μεταξύ των ε, διάφορων ε, δράσεων, ε, τα κτλ. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη αν δεν υπάρχει πρώτα ασφάλεια. Ήρθαμε σε επαφή με τους συναδέλφους από το ΕΚΟ και από την ΤΕΦΚΟ, γιατί είναι η πρώτη επιτόπου και δεν περιμένουν την ασφάλεια. Όμως η ασφάλεια θα τους βοηθήσει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Ο συντονισμός όμως ε, ε, γίνεται ανάντη και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μας, απο... Ε, μας βοηθά να αποφύγουμε παραγωγικές δράσεις. Όσο ένα παράδειγμα. Τα γαλλικά στρατεύματα προσπαθούν στις συνοικίες του Μπαγκή να επιφέρουν ασφαλείς συνθήκες διαβίωση για να επανέλθουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι και να μην κατοικούν περί το αεροδρόμιο. Αν δεν είχαμε συμπαραταχθεί με τους φίλους από το ΕΚΟ θα είμαστε αντιπαραγωγικοί γιατί το ΕΚΟ βοηθούσε ανθρώπους οι οποίοι ε, συνέρεαν γύρω από το αεροδρόμιο. Υπάρχει μια μεγάλη μάζα λοιπόν κόσμου και θα μπορούσε να έχει κινητοποιηθεί και το αεροδρόμιο. Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό για τη δράση των στρατευμάτων που όμως ήθελαν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια. Και επειδή παρακολουθώ την εξέλιξη και νομίζω ε, ότι μπορούμε να ε, καταδείξουμε ότι όλα τα εργαλεία θα πρέπει να τα συντονίζουμε και να τα ε, χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα, όχι βαθμιδό. Και στο δεύτερο διαμέρισμα του μπάνκου με τις τοπικές θρησκευτικέ αρχές και τις τοπικές αρχές υπήρξε συντονισμός για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια σε, αυτά τα, σε αυτές τις συνοικίες με την παρουσία της γαλλικής επιχείρησης και της ΜΙΣΚΑ και ξεκίνησαν κάποια project από τους φίλους μας από την ΕΦΚΟ για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να υπάρξει σταθεροποίηση. Πρέπει λοιπόν να ε, καταπολεμήσουμε μια αντιπαραγωγική ε, χρήση πρέπει των μέσων που έχουμε στη θέση μας, άρα πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα. Επίσης πρέπει να εκφράσω ότι λύπη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ένωση, ότι έχει πέντε δηλαδή ε, στρατηγία. Η Κεντρική Αφρική είναι ένα παράδειγμα αυτής της συνολικής προσέγγισης για την οποία τόσο μιλάμε αλλά δεν την εφαρμόζουμε ποτέ στην πράξη, για κοινέ δράσεις μιλάμε κτλ. Αλλά αυτή τη φορά μιλάμε για συνδυασμό όλων των εργαλείων για να σώσουμε την Κεντρική Αφρική, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία δηλαδή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλό θα ήταν να είχαμε ένα στρατηγείο στις αλλά δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς αυτό. Τώρα για τις ε, ανάγκες ή μίλησα. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας. Δεν είναι πρόβλημα γαλλικό. Αν είχαμε πει ότι είναι κίνδυνος ε, το Μάλι για την Ευρώπη, για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, δεν μας έκαναν να πάμε εκεί αυτή η κίνδυνη. Αλλά έχουμε το κίνδυνο γενοκτομίας, είναι ε, η ανθρώπινη μιζέρια, η ανάφλεξη της ευρύτερη περιοχής. Ελπίζω να μην μείνουμε μόνοι μας, γιατί υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα σημαντικά, μιλάμε για εκατοντάδε ε, εκατομμύρια ευρώ για να δαπανηθούν εκεί. Υπάρχει η ευρωπαϊκή ευθύνη λοιπόν και ο συντονισμό αυτών των μέσων και έργων μα υποχρεώνει να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Και όπω είπετε, κυρία μου, η στρατιωτική επέμβαση, η γαλλική ή η ευρωπαϊκή τέλο πάντων, θα πληρωθεί από τα κράτη που θα συνεισφέρουν και όχι από του υπόλοιπου. Σε ό,τι αφορά τώρα τον μηχανισμό ε, ειρήνη, ε, το Peace Facility, το ίδιο είχε γίνει και για τη χρηματοδότηση των στρατευμάτων της ίσων για την ασφάλεια στη Σομαλία. Πρόεδρος, να δώσω σύντομα το λόγο στον κύριο Μπρόερ για το ΕΚΟ, από το ΕΚΟ μάλλον, για να μας αναφέρει την ανθρωπιστική πτυχή. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ακούσαμε μια πολύ πλήρη παρουσίαση της ανθρωπιστικής κατάστασης τη Δευτέρα στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Η παρέμβασή μου θα επιβεβαιώσει τις περισσότερες περιπτώσεις αυτά που είπαν προλαλήσαντες. Όπως είπε και η κυρία Γεωργίευα, η Επίτροπος, με κατά κάποιο τρόπο η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία δεν είναι μια λησμονημένη κρίση όπως το 2013. Η Δευτέρα λοιπόν ήταν μια σημαντική ημέρα υπό την έννοια ότι ταυτόχρονα σχεδόν είχαμε αφενός την απόφαση τη σημαντική του Συμβουλίου και από την άλλη πλευρά οι δωρητές και η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε για να επικεντρώσει τις προσπάθειές της ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την ε, προετοιμασία της ανασυγκρότησης, της ανοικοδόμησης της χώρας. Πράγματι θεωρούμε ότι όπως υπόθηκε άλλωστε πρέπει τα δύο αυτά να συμβαδίζουν, δηλαδή η ε, καθέρωση ασφάλειας, ασφαλών συνθήκων να συνοδεύεται με την ικανοποίηση των ανθρωπιστικών αναγκών και την ανασυγκρότηση, τη δημιουργία βάσεων, ε, την ανοικοδόμηση της χώρας είναι σημαντικό το περιβάλλον να γίνει ασφαλές και για την ε, διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και για να είναι δυνατή η επιστροφή των ανθρώπων, ίσως και η πρόβλεψη της αποχώρησης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Για κατανοητούς προς το παρόν λόγους υπάρχει ε, μια βούληση εκένωσης και μαζικής ε, αποχώρησης των, τσάντ, των κατοίκων Τσάντ που είναι μουσουλμανικής θρησκείας. Κοινωνική και οικονομική φορείς όμως πάρα πολύ σημαντική για την ανοικοδόμηση, για την ανασυγκρότηση της οικονομίας, φεύγουν. Αυτό είναι κακό. Και αν φεύγουν, φεύγουν γιατί δεν νιώθουν ασφαλείς. Συμφωνώ με το που είπε ο Ντιδιέ Λενουά. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό, ε, υπήρξε ε, πολύ καλό συντονισμός, αλλά με το σεβασμό της αυτονομίας των διαφόρων φορέων για τον Μπαγκή πρέπει να υπάρξει ασφάλεια, αυτό είναι σημαντικό για ανθρωπιστικούς λόγους. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την επαρχία, την Ήπεθρο. Περιμένουμε λοιπόν εκεί να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, γιατί μέχρι στιγμής μας είναι άγνωστο αυτό. Τεράστιες όμως πρέπει να είναι οι ανάγκες στην επαρχία. Και οι ανθρωπιστικέ ομάδε στα συνεργεία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές, γιατί μέχρι στιγμής δεν μπορούν να διαμείνουν εκεί. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό από ανθρωπιστικής πλευράς είναι και η πρόσβαση στο Καμέρου να είναι ασφαλής. Είναι σημαντικό γιατί μέσω εκεί δεχετεύεται η βοήθεια, ο εξοπλισμός ε, που μας είναι απαραίτητος για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό του Μπαγκή. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια παραμένει ρευστότατη όπως ακούσατε και από άλλους ο κύριος Βέστκοτ ε, το επενθύμισε ότι τις τελευταίες ώρες ε, υπήρξαν ε, συμβάντα, υπήρξαν επεισόδια με αποτέλεσμα να χάσουν 10 άτομα τουλάχιστον στην πρωτεύουσα και είναι σαφές ότι είναι πάρα πολύ λεπτό και το ζήτημα του αφοπλισμού των πρώην ανταρτών σε λέκα. Επίσης σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που θα απορρεύσουν. Πρέπει να βιαστούμε, να δράσουμε γρήγορα. Έχουν δεσμευτεί σημαντικά ποσά με την συνέλευση της Δευτέρας. 150 εκατομμύρια ανθρωπιστική βοήθεια σας υπενθυμίζω και 180 εκατομμύρια ευρώ για αναπτυξιακή βοήθεια. Και είναι σημαντικό, θα σας εξηγήσω το λόγο σύντομα, να πηγαίνουν αυτά τα δύο μαζί και να αναγγελθούν ταυτόχρονα. Θα πρέπει από εδώ και πέρα να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη εφαρμογή και τη γρήγορη εκταμείωση της βοήθειας αυτής. Από τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουμε μια διπηρεσιακή αποστολή που επιτόπου θα μας δώσει τη δυνατότητα να λάβουμε όπως με τις διάφορες αυτές ε, συνιστώσεις της οικονομικής συνδρομής της διεθνούς κοινότητας. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει καλό συντονισμός επιτόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και σε επίπεδο δωρητών και σε επίπεδο εταίρων. Πρέπει να έχουμε πολλούς εταίρους ε, καλά στελεχωμένους ε, με επαγγελματικό προσωπικό. Αναφέρθηκε και η μεγάλη ε, συμμετοχή των γιατρών χωρί σύνορα, η αντίδρασή του πριν τα Χριστούγεννα, που έχει να κάνει κυρίω με την οργάνωση και την παρουσία εταίρων αντέδρασαν. Δεν είχαν όμως τόσο πρόβλημα με τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά με την οργάνωση. Τα ποσά υπήρχαν και θα δοθούν και μεγαλύτερα ποσά. Επίσης θέματα επιμελητίας πρέπει να ρυθμιστούν, σχέτευση της βοήθειας, ε, ε, οποιασδήποτε οδούς, κυρίως βέβαια αεροπορικά και οι πτήσεις ε, εμπορευματικές, κάργο, προς τον Πανκί είναι κάτι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να γίνουν ακόμη προσπάθειες στο πεδίο του συντονισμού. Στην Κομισιόν είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε μια ανθρωπιστική παρέμβαση πλάσα. Τι θα πει αυτό. Σε πρώτο βαθμό κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά να την εντάξουμε σε μια γενική πολυδιάστατη προσπάθεια, όπως θα την χαρακτήριζα. Δηλαδή, να εξασφαλίσουμε την πληρωμή των μισθών των υπαλλήλων της κυβέρνησης. Πού θα συγκροτηθεί Τρει μήνε μένουν απλήρωτοι πάλι. Ξέρουμε ότι οι εθνοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί θα δεσμευθούν, είναι διατεθειμένοι προς αυτό, αλλά θα πρέπει και επιτόπου να δημιουργηθούν οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις για την καλή ε, ε χρήση, την χρηστή διαχείριση των πόρων. Επίση, πρέπει να ε, μπει μπρο πάλι η, οικονομία. Πρέπει να δοθούν ε, χρήματα έχουμε project υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού. Δηλαδή να δοθεί αυτή η απαραίτητη ε, οικονομική ενίσχυση για να ξεκινήσουν τοπικές αγορές. Κοινωνικές υπηρεσίες, οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να αναβαθμιστούν. Σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει ε, κοινωνική υπηρεσία σήμερα στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Η εκπαίδευση επίσης, τα σχολεία πρέπει να ξαναλειτουργήσουν, να ανοίξουν τα σχολεία. Τα παιδιά να επανέλθουν ε, σε κανονικές συνθήκες ε, φύτηση στο σχολείο. Αλλιώς μιλάμε για χαμένη γενιά. Επίσης, προσπάθειες διαμεσολάβησης ε, όχι μόνο μέσω του θρησκευτικού κινήματος αλλά και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Να έχουμε επίσης αποθέματα ε, τροφίμων, γιατί σε δύο μήνες ξεκινάει η περίοδος των βροχών και αν δεν έχουμε τις απαραίτητες ε, προϋποθέσεις για να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός ε, και να γίνει και ε, με ομαλό τρόπο η σπορά και η εσοδεία, όλη αυτή η περίοδος να αξιοποιηθεί, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα με τα αποθέματα τροφίμων για τη χώρα αυτή πολύ πρόθεσμα πρέπει να γίνουν όλα. Έχουμε μεγάλο ε, πρόβλημα χρόνου ε, και υπάρχουν ε, αυτές οι προθεσμίες του ΟΗΕ, λίγη προθεσμία τέλος Μαρτίου, πρέπει να την τηρήσουμε πάση θυσία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δύο είναι οι ομιλητές. Η κυρία θέλει να Η κυρία Λέζινγκ θέλει το λόγο. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση. Καταρχήν ε, απαντήθηκε από το συνάδελφο που έφυγε. Μας είπε ότι θα χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση από το μηχανισμό Αθηνά. Το θέμα είναι ότι από τη μία υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης της επιχείρησης του Αφρικανικού Συνδέσμου της Αφρικανικής Ένωσης. Ε, αναφερόμουν στην άλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, Αναφερθήκατε σε γενοκτονία. Είναι δύσκολο κάποιος να δεχτεί αυτή τη λέξη. Πώς εκτιμάτε την κατάσταση. Πρόκειται για γενοκτονία, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Και βεβαίως έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος μας χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη με άλλο τρόπο. Τι ακριβώς εννοείται. Όταν λέτε ναι πρόκειται για γενοκτονία ή όχι δεν πρόκειται για γενοκτονία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Και δεύτερη ερώτηση που αφορά τον εκπρόσωπο της ΕΚΟ, η επαρχία. Δεν υπάρχει πρόσβαση στην επαρχία, κατάλαβα. Αναρωτιέμαι λοιπόν με τις ε, τα στρατεύματα τα ευρωπαϊκά που θα ενδυναμώσουν αυτήν την επιχείρηση, θα έχετε δυνατότητα να ελέγξετε και την επαρχία, δηλαδή ένα μεγαλύτερο μέρος αυτής της χώρας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέσκοτ και κατόπιν στον ταξίαρχο για να μας απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Αυτό που ακούμε εδώ και καιρό είναι ότι υπάρχει κίνδυνος γενοκτονίας και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να επιταχύνουμε τη δράση. Αλλά βεβαίως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μία διαφορά, μία διάκριση μεταξύ της εθνοκάθαρσης και του, της γενοκτονίας. Οι δύο λέξεις δεν είναι ταυτόσιμες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όταν κάποιος χωρίζει τις κοινότητες και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί ουσιαστικά δημιουργούμε δύο διαφορετικές κοινωνίες. Αλλά η μεγάλη προτεραιότητα βεβαίως είναι η συμφιλίωση πριν τη συμφιλίωση πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Σίγουρα δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση. Και εκεί οδήγησαν, αυτά οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που πραγματικά μας εντυπωσίασε μιλώντας για με πολλούς εκπροσώπους της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας είναι ότι πραγματικά εμάς δεν μας χαρακτηρίζει αυτό. Δεν αναγνωρίζουμε αυτή την κατάσταση γιατί επί πολλά χρόνια ζήσαμε ειρηνικά, συνεπάρξαμε μεταξύ των κοινοτήτων, δηλαδή δεν υπήρχε ένταση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει αντίθεση με αυτό που είπε ο πρέσβης. Εγώ Βεβαίως μίλησα για κίνδυνο, κίνδυνο γενοκτονίας, ευαίσθητη κατάσταση και μιλάμε ουσιαστικά για τους πρώην Σελέκα λέγοντας ότι θέλουμε να τους αφοπλίσουμε και να μην έχουν βαρύ οπλισμό. Λέγαμε επίσης ότι όσο δεν υπάρχει ασφάλεια στην πόλη του Μπάγκη δεν μπορούμε να επεκταθούμε και να πάμε αλλού στην επαρχία. Όταν μιλούσαμε για τις δυνάμεις του Τσάντ, τους μουσουλμάνους, αυτό που λέγαμε είναι ότι η ατιμορρησία, η αναρχία, η έλλειψη ελέγχου μπορεί, και αυτό το είδαμε σε άλλες χώρες της Αφρικής, να δημιουργήσει τις προϋποθέτης για γενοκτονία. Υπάρχει ο κίνδυνος, υπάρχει αν θέλετε η ευαισθησία και το περιβάλλον το οποίο αν δεν το ελέγξουμε και αν δεν φτάσουμε σε αυτήν την συμφιλίωση, κινδυνεύει να υπάρξει γενοκτονία. Δεν είναι αντιφατικό με αυτό που είπε ο πρέσβης. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφόρηση. Εμείς θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση επιτόπου και όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά την ανθρωπιστική πτυχή και η δική μας, αν θέλετε, υποεπιτροπή θα παρακολουθήσει ιδιαίτερα την επιχειρηση UFOR στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο για τις επιτόπου δυνάμεις πώς θα δημιουργηθεί η επιχείρηση. Σήμερα αναφερό, αναφερθήκαμε στον αριθμό των 500 επιπλέον ανδρών, αλλά καταλαβαίνω ότι σήμερα ακόμα βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις, σε συζητήσεις και ελπίζω σύντομα να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον ταξίαρχο και θα περάσουμε τώρα, κύριε Πρέσβη, στο νότιο Σουδάνα. Νότιο Σουδάν. Νομίζω όλοι γνωρίζετε ότι εδώ πρόκειται για μια κατάσταση έκρηκνη μετά τα τέλη του 2013 δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται και εδώ δεν έχουμε ακριβώς αποστολή ε, πολιτικής ασφαλείας και άμυνας υπήρχε μια επιχειρήση που ολοκληρώθηκε στη Ζούμπα. Δεν νομίζω ότι ήταν και λανθασμένη η κίνηση εκείνη και δεν είχαμε προλάβει να δούμε καν τις λεπτομέρειες της, αλλά δεν νομίζω να στενοχωριέται κονίζει γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε κυρίως για πολιτικές προσπάθειες με ειδικού απεσταλμένους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Κέρα της Αφρικής, και τις ανθρωπιστικές ε, διαστάσεις που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Westcott να μας ενημερώσει και πάλι για τα θέματα αυτό, αλλά και τον κύριο Βάουερ από την ε, ΕΚΟ και την συνάδελφο κυρία Κρυτού από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Κρητού. Ευχαριστώ πολύ. Ως Επιτροπή Ανάπτυξης ανησυχούμε ιδιαίτερως για την ανθρωπιστική διάσταση του Νοτιού Σουδάν που τόσο γρήγορα επιδεινώνεται. Σε αντίθεση με όσα είπαμε για την κεντροαφρικανική δημοκρατία, δεν μπορεί να πει κανεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η διεθνή κοινότητα συνολικά έχουν παραμελήσει το Νότιο Σουδάν τα τελευταία χρόνια. Το 2011 και 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μια σειρά από προγράμματα με αξία 185 και 185 εκατομμύρια ευρώ ε, αντιστοίχως για την εκπαίδευση, την παιδεία, την υγεία και το κράτος δικαίου. Κάποια προγράμματα ολοκληρώθηκαν πέρσι και η Επιτροπή μας, ακριβώς γι' αυτό ενέκρινε έκθεση που προετοίμασε η συνάδελφος Ντεκεζέρ για την οικοδόμηση κράτους και την ανάπτυξη στο Νότιο Σουδάν. Ήδη από την έκθεση αυτή εντοπίσαμε ότι δεν είχε κλείσει όλα τα καθήκοντα η διεθνή κοινότητα σε σχέση με τη συνολική ειρηνευτική συμφωνία του 2005 και την εφαρμογή τη. Επιπλέον, ζητήσαμε για μια επιπλέον προσπάθεια από την κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν καθώς και του διεθνεί εταίρου να προσπαθήσουν να υπάρξει εφοπλισμό και των ενόπλων παραστατικών ομάδων καθώς και να ολοκληρωθούν εσωτερικέ μεταρρυθμίσεις. Φάνηκε ότι ήταν ε, παράλογο να μην έχει ειδικό απεσταλμένο για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς τόσα παραμένουν να γίνουν. Η σημασία οικοδόμησης κράτους και ανάπτυξη θα μπορούσε να ε, φανεί εάν δεσμευτούν σε αυτά και η κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν και υπάρχει λογοδοσία με ε, συνολική διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες επικεντρώνονταν στα ανεπίλητα ζητήματα και τις εντάσεις μεταξύ βορρά και νότου της χώρας. Αυτό ήταν λογικό και απαραίτητο, όμως είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω ένταση στο Νότιο Σουδάν και δεν είχαμε δώσει αρκετή προσοχή σε αυτό το στοιχείο. Σε σχέση με την τωρινή κατάσταση στο Νότιο Σουδάν και τους ηγέτες του υπάρχουν ε, δυνατότητες υπάρχει δυστυχώς περίπτωση κλιμάκωσης και πρέπει να δοθεί τέρμα τώρα. Οι δηλώσεις του κυρίου Σαλβακύρ, οι χθεσινές, είναι πολύ ανησυχητικέ για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει κάτι να γίνει. Παρ' όλα αυτά μπορεί να ε, δίδαγμα να το αντλήσουμε από την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν και μπορεί αυτά στο μέλλον να είναι χρήσιμα και για το ίδιο το Νότιο Σουδάν αλλά και για άλλε χώρε. Για μα, στην Επιτροπή Ανάπτυξη, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι πιστεύουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ACC σε σχέση με τα προγράμματα βοήθειας που υπό τις τωρινές συνθήκες δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως. Όμως μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αν πιστεύετε ότι χρειάζεται επαναπροσανατολισμός της βοήθειάς μας μόλις υπάρξει κάποια ε, περισσότερη ειρήνευση στην περιοχή. Ευχαριστούμε κύριε Κατσού. Ο κύριος Βασκότ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα δίσταζα να περιγράψω την κατάσταση του Νότιου Σουδάν αυτή τη στιγμή ως τραγική. Ως το νεότερο έθνος του κόσμου, εγώ ε, με την κυρία Άστον παρευρεθήκαμε στους εορτασμούς της ανεξαρτησίας το 2011, έχει πέσει θύμα, όπως νέες χώρες συχνά υποφέρουν από αυτό, ε, έχει πέσει θύμα εμφύλιας σύραξης και δεν βλέπουμε να υπάρχει και προοπτική τέλους αυτό. Κάθε κίνημα ανεξαρτησίας τίνει να είναι ένας συνασπισμός. SPLM, SPLA, διαφορετικές ε, πολιτικές ε, οικογένειες. Πάντοτε ήταν ε, γνωστό ότι το SPLM αποτελείται από διαφορετικές ομάδες που συγκεντρώθηκαν για να πολεμήσουν για την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν με τη διεθνή στήριξη επίσης τα κατάφεραν και είχαμε αρκετές ελπίδες ότι η οικοδόμηση κράτους που έπρεπε να ακολουθήσει καθώς δεν υπήρχαν κρατικές υποδομές ούτε καν ε, υλικέ. αυτό θα οδηγούσε σε νέα θεσμικά όργανα με σταθερές γερές πολιτικές δομές επιπλέον με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλευρό τους για να το στηρίξει. Μόλις πρόσφατα είχε υπογραφεί μια σύμβαση για την οικοδόμηση κρατικών κτηρίων. Όμως, οι πολιτικές εντάσεις εντός του FPLM άρχισαν να καταλήγουν σε βιαιότητες. Στις 15 Δεκεμβρίου, μάλιστα, είχαμε επεισόδια στην Εκτελεστική Επιτροπή και αυτό ε, άρχισε να διαδίδεται στην υπόλοιπη χώρα και έχει οδηγήσει σε σύγκρουση, ένοπλη σύραξη μεταξύ διαφόρων αντίπαλων ομάδων. Η κατάσταση από στρατιωτική σκοπιά είναι περίπλοκη. Και παρόλο που υπάρχει μια ομάδα επαναστατών οι οποίοι μπορούν να εντοπιστούν, ε, οι οποίοι είναι πιστοί στον Αλ Μασάρ, τον πρώην αντιπρόεδρο, ενώ υπάρχουν πολλοί κρατούμενοι, περίπου 12 πολιτικοί τους οποίους κρατά η κυβέρνηση στην Τζούμπα, διαφορετικών προελεύσεων, Ντίγκα, Ενούρα, δεν είναι όλοι της ίδιας ομάδας στη χώρα, αλλά παρά τις εκκλήσεις μας για την απελευθέρωσή τους, παραμένουν σε κάθριξη, στη φυλακή. Ε, η κατάσταση συνεχίζει να ε, υποβαθμίζεται, να επιδεινώνεται. Ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 10.000 έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους αυτή τη σύγκρουση. Περίπου μισό εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί. Κάποιοι ε, μία και δύο φορές. Κάποιοι δραπετεύουν από τον Νότιο Σουδάν στο Σουδάν για να γλιτώσουν. Το αντίστροφο από το που συνεβαίνει προηγουμένως. Και όσο πιο πολύ κρατάνε οι εχθροπραξίες, και εδώ, όπω και στην κέντρο-αφρικανική δημοκρατία, μπορεί οι εθνοτικές διαφορέ να γίνουν ακόμη πιο βαθίε και η κρατική δομή να καταρρεύσει. Τι γίνεται λοιπόν για να επιληθεί η κατάσταση. Την ηγεσία έχει αναλάβει η IGAD, στην οποία προεδρεύει η Αιθιοπία, ο περιφερειακός οργανισμός, η οποία προσπαθεί να προβλέψει μια διαδικασία διαιτησίας Ένας ε, πας ε, διαιτητής έχει οριστεί για τη διαδικασία αυτή με συμμετοχή της Ουγκάντα, της, ε, του Σουδάν και της Κένια. Ε, έχουν πάει στην ε, Τζούμπα προσπαθώντας να προσπάσουν την απελευθέρωση των κρατουμένων, να συζητήσουν με τον πρόεδρο, να ζητήσουν την ε, πάυση των εχθροπραξιών και να αρχίσει και πάλι να υπάρχει μια πολιτική ζωή ομαλότερη στη χώρα, ε, μήπως λυθούν τα προβλήματα ε, ειρηνικά. Οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν οδηγήσει ακόμα σε πάυση πυρός. Ο πρόεδρος Κία είπε ότι αρχικά ήθελε να ε, υπογράψει την ε, Κεχηρία. Ο Μασάρ δεν το δέχτηκε ποτέ αυτό. Τη Δευτέρα και την Τρίτη υπήρξαν ε, συνομιλίες και προβλεπόταν σύνοδο της Άγκατ στην Τζούμπα σήμερα. Όμως αναβλήθηκε η συνάντηση η σημερινή. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Και πραγματικά προσπαθούμε να έχουμε πολιτικές εξελίξεις μαζί με την απελευθέρωση των εκδοτουμένων. Αλλά προ στιγμήν και η κυβερνητική και η πλευρά, και η πλευρά των επαναστατών θεωρούν ότι τα συμφέροντα του μεν και των δε εξυπηρετούνται καλύτερα με την ένοπλη αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση πρόσφατα κατάφερε να πάρει τον έλεγχο των ε, δύο κρατηδίων ε, που είναι κατεξοχήν παραγωγή πετρελαίου στη χώρα, αλλά δεν έχει τον έλεγχο εκτός των πρωτεύουσών των κρατηδίων αυτών. Ελέγχουν λόγω χάρη την ε, πρωτεύουσα του Γιόγκλα ενός άλλου κρατηδίου, αλλά όχι το υπόλοιπο κρατήδιο. Το ίδιο και στο Unity και σε ένα ακόμη κρατήδιο του Βορρά. Η Ουγκάντα επηρεάζεται από τις εχθροπραξίες επίσης και λέει ότι στηρίζει την εκλεγμένη κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της από τους επαναστάτες που προσπαθούν να υπονομεύσουν την κρατική δομή. Αυτή είναι η θέση τους. Αυτό όμως δεν επιταχύνει την ερνευτική διαδικασία. Γιατί η επίλυση του προβλήματο αυτή τη στιγμή επιζητάται μόνο με στρατιωτικά μέσα. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε συζητήσει. Η ΆΙΚΑΤ έχει αναλάβει την ηγεσία ε, με τη στήριξη τη Αφρικανική Ένωση. Η κυρία ε, Νούα ε, επισκέφθηκε η ίδια ως πρόεδρος τη Αφρικανικής Ένωσης την περιοχή Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με την Νορβηγία, το ΝΑΤΟ και το ΟΗΕ προσπαθούν να έχουν ε, τη δική τους, ε, το δικό τους ρόλο και ο δικός μας απεσταλμένος αυτή τη στιγμή θα ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ, αλλά είναι στο κέρας της Αφρικής κάνοντας ε, το ε, μετακινούμενο συνεχώς μεταξύ Τζούμπα και το επιτελείο μας εκεί για να προσπαθήσουμε, των γραφείων μάλλον εκεί, για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα τον συναντήσω και εγώ στο χώρο δράση του. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια πολιτική λύση και η εκχειρία παραμένει πλέον άμεση ανάγκη. Οι ανθρωπιστικές ανάγκες φυσικά διαρκώς αυξάνονται θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεμπράουερ για να σα τα εξηγήσει, να σα πει καλύτερα τι κάνουμε για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό. Αλλά υπάρχουν επί τη ουσία προσπάθειε και το να υπάρξει πρόσβαση στι ομάδε των εκτοπισμένων σε όσου έχουν προβλήματα είναι πάντα δύσκολο σε ένα κράτο που βρίσκεται σε κατάσταση εμπόλεμη. Το να πάψει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Μέρο των συνεπειών τώρα αυτή τη σύγκρουση και του γεγονότος ότι γίνεται διεθνωτική και πολύ άγρια είναι ότι υπάρχουν διαρκώς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με δολοφονίες, άγριες δολοφονίες, εξοδικαστικές δολοφονίες, βασανιστήρια και το καθεξής. Η ΟΗΕ θα ετοιμάσει, θα συστήσει γρήγορα μια εξεταστική ανακριτική επιτροπή που η Αφρικανική Ένωση ελπίζουμε να στηρίξει, ώστε οι παραβιάσεις αυτές να μην καλύπτονται άλλο από ετοιμορρυσία. Ήδη θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επί του θέματος από την επόμενη εβδομάδα. Α, πρόεδρε, έγινε μια παρατηρήση για τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ έχει αναλάβει πλήρως τον ρόλο του σε αυτή την κρίση, προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες των χιλιάδων εκτοπισμένων οι οποίοι έχουν καταφύγει στα, στα, στις περιοχές που ελέγχει ο ΙΕ ο οποίος προσπαθεί να τους παράσχει μια προστασία και αισθάνονται ασφαλείς η προσφορά καταφυγίου ε, ε, καταφυγίου σε όσους έχουν ανάγκη από τον ΟΗΕ έχει οδηγήσει και σε εντάσεις γιατί η αντιπολίτευση σε αντίθεση με όποιον, ε, σε αντίθεση με όποιον έχει την εξουσία, είναι κάτι που θεωρείται αρνητικό. Ο πρόεδρος Κία έχει τοποθετηθεί αρνητικά σε σχέση με την ε, δράση του ΟΙΕ, αλλά παραμένει απαραίτητη εκεί η παρουσία τους. Επίσης για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Δευτέρας. Και εκεί αναφέρεται ότι εάν εντοπιστούν υπεύθυνοι της παρεμπόδισης της ειρηνευτικής διαδικασίας θα πρέπει να αναλυθούν μέτρα εναντίον τους. Αλλά θα πρέπει να επιδιώξουμε και συνεργασία με τις χώρες της ε, ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και της Αφρικανικής Ένωσης και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να πάψει αυτή η εκρηθμός κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Ο κύριος δεν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, αλλά για να συμπληρώσω αυτήν την παρουσίαση, μας είπε αρχικά ο κύριος Βέσκοτ ότι ήταν μια νέα χώρα και μια ευαίσθητη χώρα το Νότιο Σουδάν. Πριν ξεκινήσει η κρίση, η κατάσταση ανθρωπιστική στη Νότιο Σουδάν ήταν ήδη ανησυχητική, πολύ ανησυχητική. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με τους εκτιμήσεις 4.400.000 άνθρωποι, περίπου το 1 τρίτο δηλαδή του πληθυσμού, χρειαζόταν ανθρωπιστική βοήθεια. 3 εκατομμύρια περίπου βρισκόταν σε κατάσταση προβληματική όσον αφορά τη διατροφή τους και ήδη 230 230.000 άνθρωποι ήταν πρόσφυγες στην Αιθιοπία, στην Δημοκρατία του Κονγκό και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Όλα αυτά πριν ξεκινήσουν οι βιαιότητες και η κρίση σημερινή. Η ανθρωπιστική κατάσταση, αν θέλετε, καθημερινά γίνονται όλο και πιο ανησυχητικοί. Έχουμε κάποιες πολύ μερικές εκτιμήσεις βεβαίως, αλλά βλέπουμε ότι 560.000 άνθρωποι έχουν μετατοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, επιπλέον αυτών που προανέφερα που είναι πρόσφυγες εκτός και 110.000 πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες, κυρίως στην Αιθιοπία και στην Ουγκάντα. Τα στοιχεία αυτά βεβαίως δεν είναι στάσιμα, διαρκώς αυξάνονται και είναι, αν θέλετε, πιο ανησυχητικά τα στοιχεία σήμερα από ό,τι ήταν τη Δευτέρα όταν έγινε η παρουσίαση στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Σε σχέση λοιπόν με αυτήν την επιδίνωση, την καθημερινή επιδίνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης έχουν προβλήματα χρηματοδότησης. Ναι, όντως είχαμε προβλέψει αρχικά μια χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων για την ανθρωπιστική βοήθεια για τον Νότιο Σουδάν το 2014. Όμως, αυτά τα 50 εκατομμύρια θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για μια κατάσταση πριν την κρίση. Σήμερα, σήμερα βλέπουμε ότι πρέπει να ξαναδούμε, να ξαναεκτιμήσουμε αυτήν την επίγουσα ανάγκη η οποία διαρκώς επιδεινώνεται. Σας μίλησα για τους αριθμούς των προσφύγων που επίσης αυξάνονται, οι πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες. Πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τους μετατοπιστέντες και τους πρόσφυγες σε όλο το αφρικανικό κέρας που ήδη ήταν κρίσιμη και ε, για, αυτήν την, για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης χρηματοδότηση είναι ανεπαρκής και αυτό πριν ξεκινήσει η κρίση. Έχουμε βεβαίως προβλήματα πρόσβασης. Οι μάχες συνεχίζονται. Η κατάσταση είναι προβληματική όσον αφορά τη σταθερότητα και την ασφάλεια, αλλά και πριν την κρίση και πριν τα Χριστούγεννα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και σήμερα βλέπουμε ότι το προσωπικό όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια παρέμειναν επιτόπου. Καταφέραμε δηλαδή να έχουμε μία σχετικά ικανοποιητική πρόσβαση στις πιο επικίνδυνες περιοχές. Παρά όλα αυτά, η κατάσταση δεν είναι σταθερή, όπως σας είπα. Ο πρόεδρος Κύρ πριν από δύο ημέρες αναφέρθηκε με πολύ επιθετικό τρόπο κατά του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και, και αυτό μπορεί να εξηγηθεί, κατά των ανθρωπιστικών οργανισμών. Οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας. Βεβαίως εμείς εδώ Συνεργαζόμαστε στενά με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και βεβαίως θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να συνδέσουμε την πρόσβαση με το θέμα της εκεχηρίας. Η ανθρωπιστική πρόσβαση είναι κάτι που πρέπει σαφώς να το δούμε ανεξάρτητα και όπως είπε και ο κύριος Βέσκοτ, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για να απομακρύνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Τι προκλήσεις έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να είναι στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών. Να έχουμε πρόσβαση, να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και όπως έγινε και στην κεντροαφρικανική δημοκρατία, θα πρέπει να φτάσουμε το επίπεδο 3 και για τον Νότιο Σουδάν όσον αφορά τον χαρακτηρισμό του επίγοντος χαρακτήρα της ε, κατάστασης επιτόπου. Κινητοποίηση κονδυλίων που να ανταποκρίνονται στην σοβαρότητα της κατάστασης. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής Ανάπτυξης. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στο θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και στον συνάδελφό μου. Ευχαριστώ, Γιάννη Λουίς. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Πολύ σύντομα να πω ότι εμείς από την πλευρά της αναπτυξιακής βοήθειας προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από κοινού βεβαίως με τα κράτη-μέλη και με άλλους σημαντικούς φορείς. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας, προηγούμενες επιχειρήσεις και βεβαίως να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει μια σειρά δράσεων και επιχειρήσεων προσπαθώντας πάντα να προσαρμοστούμε στη πραγματικότητα. Πρώτον, αναθεωρούμε τις επιχειρησιακές μας ε, δυνατότητες από τις 15 Δεκεμβρίου που είμαστε επιτόπου παρόντες. Έχουμε έρθει σε επαφή με όλους τους φορείς, μη κυβερνητικοί οργανισμοί κατά κύριο λόγο, οι οποίοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται επιτόπου σε κάποιες από τις περιπτώσεις πρέπει να διακόψουμε τη δράση μας. Οι περισσότεροι μη κυβερνητικοί οργανισμοί με του οποίου συνεργαζόμαστε μας είπαν, μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να συνεχίσουμε για την προστασία των παιδιών, των γυναικών, για θέματα στήριξης του πληθυσμού, επίσης μια πιο στρατηγική δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οθετήσει στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος του 2013, μια σειρά προγραμμάτων στο τομέα της υγείας, της ε, γεωργίας, της διατροφής, της διακυβέρνησης και της παιδείας. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την πληρωμή του εκπαιδευτικού προσωπικού στην περιοχή. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι η δράση μας εμποδίζεται από την κατάσταση επιτόπου. Θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε μια νέα στρατηγική από κοινού με τα κράτη-μέλη και τους άλλους συνεργαζόμενους φορείς, έτσι ώστε να καθορίσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες να συνεχιστούν κάποια προγράμματα ή να αναπροσαρμόσουμε κάποια άλλα. Αυτή η αναθεώρηση βεβαίως γίνεται σε στενό συντονισμό με τους συναδέλφους από την ΕΚΟ. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιοχές τις οποίες δεν μπορεί να έχει πρόσβαση η ΕΚΟ λόγω οικονομικών περιορισμών. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Μένουν ακόμη λίγα λεπτά για να γίνει μια συζήτηση. Δεν ξέρω ποιος από τους συναδέλφους θα ήθελε το λόγο. Δύο βλέπω. Ε, ο κύριος Κατσμάρεκ. Να είστε σχετικά σύντομοι, παρακαλώ, δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους κύριους καταρχά για τις παρουσιάσεις τους, για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Βέβαια, όταν μιλάμε για τον Νότιο Σουδάν, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ε, δύο βασικοί πυλώνες, το εισόδημα από τα έσοδα, μάλλον από το πετρέλαιο. Και η αντιπαράθεση, η σύγκρουση, γιατί ξέρουμε ότι όποιος κερδίσει θα ωφεληθεί. Ε, επίσης, ε, πρόβλημα είναι πού οφείλεται αυτή η αντιπαράθεση. Είναι εθνοτική λόγη, είναι το πετρέλαιο. Εάν δεν διαγνώσουμε καλά την κατάσταση, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λάβουμε και την κατάλληλη και την σωστή απόφαση η Ουγγάντα. Φυσικά και δεν μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει από τη μία τον πρόεδρο και από την άλλη να προσπάθει να κάνει το μεσολαβητή. Δεν μπορείς να είσαι με το ένα πόδι από τη μία πλευρά του φράχτη και με το άλλο από την άλλη. Και πρέπει να γίνονται λεπτές οι ρίζες, οι αιτίε του προβλήματος. Μήπως είναι η Κίνα η βασική πελάτης ε, πετρελαίου από το Σουδάν. Τι ξέρουμε λοιπόν για την Κίνα, τι κάνει η Κίνα θεωρητικά θεωρητικά τουλάχιστον επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ενδιαφέρει εκείνο να τερματιστεί αυτή η αντιπαράθεση για να έχει πάλι πρόσβαση στο πετρέλαιο. Κυρία Λέζινγκ το έχει το λόγο. Ναι. Είπατε ότι θέλετε να εμπνευστείτε και να βασιστείτε στην παρελθούσα εμπειρία σας. Το θέμα είναι αν κάποια από τα σφάλματα που κάναμε στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, με διεθνή στήριξη βέβαια, πολλές φορές οδήγησε σε διάσπαση κάποιων ε, χωρών. Τι μπορούμε εδώ να κάνουμε καλύτερα και πολύ συγκεκριμένα θα ήθελα να σας ρωτήσω. το θέμα των αστυνομικών δυνάμεων και των ενόπλων δυνάμεων του Νοτιού Σουδάν. Τι μπορεί να κάνει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει την ανασυγκρότηση αυτού του κράτους. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρος. Υπάρχουν άλλα σχόλια, παρατηρήσεις. Όχι. Επομένως, θα δώσω ε, στους δύο κυρίους το λόγο. Ο κύριος Westcott, καταρχάς. Ευχαριστώ. Τι ε, είναι αυτή η σύγκρουση που οφείλεται. Φυσικά πολλές φορές το αίτιο είναι η φυσική πόρη και άλλα πράγματα βέβαια και σίγουρα ε, έχει να κάνει και με τη διάσπαση της συμμαχίας του ενώ ο πρόεδρος Κία απέλησε ε, υπουργούς, έδιωξε υπουργούς τον Ιούλιο οπότε αυτοί πλέον δεν ήταν μέλη της κυβέρνησης και δεν είχαν πρόσβαση στις ε, αποφάσεις για τη διανομή των πόρων και είμαι βέβαιος ότι και αυτό συνεισέφερε στην ε, διάσπαση της όλης αυτής ε, διαδικασίας. Τώρα, για τον Νότιο Σουδάν είναι μια φτωχή, ευάλωτη, έφραστη χώρα με μεγάλα πετρελικά αποθέματα που έρχονται ως ρευστό. Άρα μία από τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία της ανασυγκρότησης είναι να βελτιωθεί η διαδικασία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο της κυβέρνησης. Εκεί παρέχουμε εμείς ε, στήριξη στην ε, νοτιοσουδανική κυβέρνηση. Πριν όμως ε, ομαλοποιηθούν τα προγράμματα παροχή βοήθεια προ την κυβέρνηση, θα πρέπει να έχουμε ορατή βελτίωση σε αυτή τη χρηματοοικονομική διαχείριση, να υπάρχει διαφάνεια, κυρίως για τον κόσμο, του κατοικού του Νότιου Σουδάν και βέβαια και για την διεθνή κοινότητα σε δεύτερη φάση. Ο ρόλο τη Κίνα, καλή ερώτηση. Φυσικά και ε, ενδιαφέρεται και για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Διπλωματικά έχουν δραστηριοποιηθεί οι Κινέζοι, έχουν υποστηρίξει τη διαδικασία διαμεσολάβησης Ίσως θα έπρεπε να είχα αναφέρει την Κίνη γιατί έχουμε επαφή και αυτοί κρατάνε επαφή μαζί μας, ε, στο χαρτούν, έχουν πρόσβαση και ένα από τα περίεργα αυτής της σύγκρουση είναι ότι το Σουδάν δεν έχει τοποθετηθεί, δεν έχει πάρει την πλευρά καθενός, ε, δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση και αυτό είναι καλό. Η κινέζικη επιρροή, επομένως, μπορεί και να μην είναι άσχετη με αυτό το γεγονός. Πάντως όλη η διεθνής κοινότητα εργάζεται και δεν βλέπω να διαφοροποιούνται απόψεις μεταξύ των μέλων. Τώρα για την ΕΓΚΑΤ, αυτή τη διαδικασία μεσολάβησης, ε, η Αιθιοπία που προεδρεύει ε, διευθύνει με πολύ μεγάλη μαϊστρία της ε, διαπραγματεύσεις. Αν ήταν η διχοτόμηση του Σουδάν λάθος, και ανεξάρτηση του Νοτιού Σουδάνου. Ξέρετε, με αυτό τέλειωσε ένα 20 εμφύλιος. Και από αυτές τις συνθήκες δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να επιληθεί ε, το πρόβλημα και οι πολιτικές δυσκολίες που είχαν ανακύψει. Βέβαια, όλοι και στην περιοχή και στη διεθνή κοινότητα ανησυχούν μήπως υπάρξει περαιτέρω ε, κατακαιρματισμό στο Σουδάν, δηλαδή με μια διχοτόμηση και του Νότιου Σουδάν. Το θέμα είναι να μπορούν ε, οι πολίτες να διευθετούν τις διαφορές τους χωρίς ε, να προσφεύγουν στην βία. Γι' αυτό και στόχος της ΆΙΚΑΤ είναι και δικός μας. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ε, στερεές ε, πολιτικές δομές στο Νότιο Σουδάν. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω ποιος θέλει, ο κύριος Γκαρίγα, ο κύριος Ντεμπόρ και οι δύο. Κανείς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε και το σημείο αυτό της μερισιάς διάταξης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους μας τους προσκεκλημένους και τους συναδέλφους μας βέβαια. Μπορείτε να παραμείνετε αν θέλετε για τη συζήτηση της αντιπυραυλικής άμυνας βέβαια, έτσι. Οι συνάδελφοι λοιπόν των Επιτροπών Εξωτερικών και Ανάπτυξης. Πάντως σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Okay, uh, Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση σαν ποτέρχο για την αντιπυραυλική ασπίδα. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περιμένω απλώς να βάλουν να φύγουν όσοι δεν έχουν ε, ενδιαφέρον για τη συζήτηση από την αίθουσα. για ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί σκιώδεις, να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλια που έχετε υποβάλει ως τώρα και για τις τροπολογίες σας. Ε, ευθύς εξ αρχής ήταν σαφές ότι η έκθεση αυτή θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω του θέματος. Διαφορετικές απόψεις ακούστηκαν και η πρώτη ανάγνωση το επιβεβαίωσε. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση των σχεδόν εισηγητών όπου προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις απόψεις των διαφορετικών ομάδων. Και είδαμε και σε εκείνη τη συνάντηση και σε προηγούμενες ότι δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συνένεση. Στο επίπεδο της Επιτροπής μας, κάτι που το ανέφερα και στο προηγούμενο σχέδιο. Όμως είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να ετοιμάσει την έκθεση αυτή τελικά, να την ε, συντάξει και να εγκριθεί και σε αυτή την ε, θητεία. Γι' αυτό θα έλεγα να Πάμε ένα βήμα πίσω για να μπορέσουμε στη συνέχεια να πάμε δύο βήματα μπροστά. Θα χρειαστώ λοιπόν επιπλέον χρόνο, επιπλέον χρόνο για να συντάξω με, ένα νέο ακριβέστερο κείμενο διότι δεν είναι απλό να έχουμε για ένα τόσο ευρύ θέμα συμφωνία. Υπάρχουν πάντως σημεία στα οποία μπορούμε να επιτύχουμε ε, κάποια βαθμό σύγκλησης δεν σημαίνει ότι η έκθεση θα αναβληθεί επάπειρον, απλώς θα μπορέσουμε να την βελτιώσουμε ελπίζω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και παρακαλώ να μου δώσετε τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Τερχό. Ε, είμαι σε κάπως ιδιαίτερη θέση γιατί θα πρέπει να δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Προεδρεύω στη συνεδρίαση αλλά είμαι και σχεδόν εισηγητές εκ μέρους του ΕΛΚ. Για να είμαι ακριβέστερος θα μιλήσω πολωνικά. Proszę Κυρίες και κύριοι, είμαι σε κάπως άβολη θέση, διότι επανειλημμένως σε διάφορες συναντήσεις μου ζητήθηκε από τον Δ. Πάσκου και την κυρία Νικολάη, τους υπόλοιπους εισηγητές των Σοσιαλιστών Δημοκρατών και της Άλντε, να παρουσιάσω την κοινή μας θέση για την έκθεση αυτή. Να πω ότι συμφωνώ απολύτως με όσα είπε ο κύριος Τέρχος, ε, συζητητής. Το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Είναι αμφιλεγόμενο. Και κατά κάποιο τρόπο, κατά μία έννοια, δεν είναι απλώς θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που αρχίσαμε να περιλαμβάνουμε στην έκθεση Δηλαδή η ιδέα, οι δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχοληθούν με την αντιπυραυλική ασπίδα της Ευρώπης είναι κάτι που ως τώρα δεν υπήρχε. Είναι ένα καινούριο τελείως σχέδιο. Κανένα από τα κράτη-μέλη δεν έχει αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από οργανωτικής και οικονομικής σκοπιάς μια αντιπυραυλική ασπίδα. Στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν τουλάχιστον προς αυτό. δεν θέλουμε να ε, έρθουμε και να επαναλάβουμε προσπάθειες του ΝΑΤΟ. ένα οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν και τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα όπως ε, το έχουν ε, εφαρμόσει ως τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Μιλάμε για ένα αμερικανικό σύστημα που σε διμερή βάση έχει δημιουργηθεί σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως θα πρέπει να συμπληρώσει τη δράση του ΝΑΤΟ ώστε να προστατεύονται όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο όσοι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη Σύνοδο του Σικάγο όλοι συμφώνησαν σε αυτό. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα που τα ερχόμενα χρόνια δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί, μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Ε, εάν υπάρχει στενή συνεργασία ε, εμβαθυμένη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ σε σχέση με αυτό το θέμα μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές εξελίξεις. Ο κύριος Πασκού λοιπόν και η κυρία Νικολάη μου ζήτησε να σας πω ότι ως και όδης εισηγητές και εκ μέρους των τριών πολιτικών ομάδων στηρίζουμε την ιδέα επανασύνταξης του κειμένου στο δυνατόν συντομότερα για να είναι ακριβέστερο και να μην περιλαμβάνει τόσες πολλές ιδέες, να μην καλύπτει τόσο διαφορετικά ζητήματα που μπορεί να είναι αμφιλεγόμενα και που να μην επιτρέπουν τη συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Πάντως, ε, δεχόμαστε το εξής. Δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε την ασφάλεια των κρατών μελών. Και εάν είναι απαραίτητο, θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο τα μέλη του ΝΑΤΟ, να προστατεύονται από μια αντιπυραυλική ασπίδα εφόσον δημιουργηθεί στο μέλλον. Οι τρει μα λοιπόν, μετά την χθεσινή συνάντηση των Σκιωδών, έχουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε σκληρά τι ερχόμενε ημέρε, προκειμένου να επανασυνταχθεί εγκαίρω το κείμενο. Ε, είμαι βεβαίω ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε ένα νέο σχέδιο κειμένου, ένα νέο σχέδιο έκθεση, μέσα σε λίγε ημέρε σε συνεργασία με τον εισηγητή και για να αποφύγουμε εκατοντάδε νέε τροπολογίε που θα μπορούσαν να υποβληθούν. Διότι εάν συνεργαστούν τουλάχιστον τέσσερι πολιτικέ ομάδε, ελπίζουμε ότι η όλη διαδικασία θα γίνει πολύ πιο ε, γοργή. Υπάρχουν σχόλια από τους συναδέλφους. Όχι. Κύριε Τέρχο, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι σε συνεργασία με τη Γραμματεία για τις προθεσμίες υποβολής τροπολογιών μπορούμε να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το νέο κείμενο αμέσως. Ευχαριστούμε πολύ και θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Πολύ ωραία. Με χαρά μου τώρα να υποδεχτώ τους νέους μας καλεσμένους. Τον ε, Μάβαρχο nobody is perfect. Um, Director Concepts and Capabilities EU staff, EU military staff, who is replacing Admiral Williams, who sent his apologies. Mr. Giorgio. Να υποδεχτώ τον κύριο Williams, να υποδεχτώ. Management and Planning Directorate. Τους συμμετέχοντες, τον κύριο Hans Bernhard Weissert, που είναι υπεύθυνο του Ευρωπαϊκή ε, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για την Ασφάλεια και την Άμυνα, τον κύριο, τον κύριο Πόρτζο και τον κύριο Μπρουσ Βίλιαμς. Θα συζητήσουμε για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Ευρωκοινοβούλιο, διότι έχει γίνει πολλή συζήτηση ως τώρα και γνωρίζουμε πόσο ουσιαστικό είναι το πρόβλημα της σωστής εκπαίδευσης των στρατιωτών, του στρατιωτικού μας ε, δυναμικού. Για τα θέματα λοιπόν εκπαίδευσης να δώσω το λόγο στον ε, στρατηγό Λερού. Θα σας παρακαλέσω να παραμείνετε σε μια εισήγηση των 6-7 λεπτών, 10 το πολύ, για να έχουμε χρόνο και για διάλογο. Έχετε το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συντομεύσω, όπως μου ζητήσατε. Θα είμαι πολύ περιεκτικός, ώστε και οι συνάδελφοί μου που επίσης εργάζονται στον τομέα αυτό να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο, γιατί είναι ομαδική δουλειά που κάνουμε. Έχετε λοιπόν μπροστά σας ε, ένα μέρος, μια ε, μερίδα της ομάδας αυτής. Ουσιαστικά θέλουμε να έχουμε μια, ένα απόθεμα στρατιωτικών δυνάμεων. Συμμετέχουν πολλοί παράγοντες και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αυτών των φορέων. Μιλήσαμε διαμακρών σήμερα για το πώς μπορεί συγκεκριμένα να γίνει πιο ορατή η στρατιωτική δράση. Αυτό αποτελεί καρπό προκατακτικής δουλειάς, μέρος της οποίας βέβαια είναι η επιμόρφωση, η κατάρτιση. Πώς λοιπόν ε, βλέπουμε την κατάρτιση, την εκπαίδευση ε, και στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης, ε, της μείωσης των προϋπολογισμών. Φυσικά θέλουμε να δημιουργήσουμε δυνατότητες σχετικές και εκεί ο άνθρωπος, η κατάρτιση η εκπαίδευσή του έχει ένα κεντρικό ρόλο. Και αυτή είναι η σημασία της ανάπτυξης ε, δυνατοτήτων ε, της εκπαίδευσης ε, της κατάρτισης. Θα σας παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα λοιπόν τα πράγματα. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες της παρεμβασής μου. Πρώτος, ανάπτυξη δυνατοτήτων, μίλησα γι' αυτό. Δεύτερον, πρόθεση μιας κουλτούρας ασφάλειας και άμυνας, κάτι σημαντικό. Και τρίτο, Λίγο πολύ κάτι που συζητήσατε με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αυτό κάνουμε και εμείς στο Μάλκι και στη Σομαλία. Σήμερα δηλαδή εκπαίδευση μονάδων ε, στρατιωτικών δυνάμεων από τρίτες χώρες ή τρίτες οργανώσεις. Αυτό το ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκπαίδευση, θέλουμε να ενταχθεί στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων. Σήμερα δουλεύουμε πάνω ε, στα στρατηγία μας και στην εκπαίδευση των μελών των στρατηγίων. Η τακτική είναι ένας βασικός άξονας, ε, όχι ο μόνος βέβαια. Βλέπουμε επίσης ότι η εκπαίδευση στα στρατηγία ε, και τον, ε, η εκπαίδευση των ε, τακτικών σχηματισμών είναι ένα σημαντικό εργαλείο και είναι και ένα πεδίο πειραματισμού θα το χαρακτήριζα για να σε δούμε συγκεκριμένα και να αποκρισταλώσουμε εμπειρίες στον τομέα της εκπαίδευσης της άσκησης των στρατιωτών μας και του προσωπικού μας. Επίσης βλέπουμε ότι είναι και ένα πεδίο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που χαρακτηρίζεται ήδη σε κάποιες ε, μονάδες ε, έχουμε ε, την ενάερια μονάδα μεταφορών που είναι ένα παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρεται σε ό,τι αφορά την κοινή χρήση και συγκέντρωση πόρων, το pooling and sharing δηλαδή. Αυτό το pooling and sharing εφαρμόζεται πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ σωστό τρόπο στον τομέα της εκπαίδευσης της κατάρτισης. Και εκεί δίνουμε έμφαση και στο επίπεδο του στρατηγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλα νέα πεδία δράσης που αναδεικνύονται και τα οποία αναφέρει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπέρασματά του, όπου θα πρέπει δηλαδή να καταβάλουμε σίγουρα προσπάθειες. Ο κυβερνοχώρος, σίγουρα, η θαλάσσια ασφάλεια, διαχείριση των συνόρων, ενεργειακή ασφάλεια. Αυτά είναι ορισμένα από τα πεδία δράσης όπου πολύ ε, σίγουρα έχουμε δυνατότητε πρόοδου και να καινοτο, μπορούμε να καινοτομήσουμε. Επίσης, συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη και τα έθνη, τα 22 τουλάχιστον, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους σε επιχειρήσεις της Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, ε, σε συμμαχίες ή ε, ως κράτος έθνος. Και βέβαια θα πρέπει να μπορεί το στρατιωτικό σκέλος να ε, επέμβει, έχοντας δηλαδή εκ των προτέρων την εκπαίδευση και την κατάρτιση για να φέρει σε πέρα στα καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Πρόθεση λοιπόν, δεύτερο σημείο, μιας κουλτούρας, πώς να το πω, μιας νοοτροπίας για την ασφάλεια και την άμυνα. Μιας ευρωπαϊκής τέτοιας κουλτούρας. Το πρώτο σημείο εφαρμογή που βλέπω, ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγουμε, θα έλεγα σχεδόν αμυγός στρατιωτικά υβρύτερα. ευρύτερα στο πλαίσιο μια γενική ε, συνολική προσέγγιση με του διπλωμάτε φίλου μα και όλου του μη στρατιωτικού παράγοντες με του οποίου συνεργαζόμαστε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτή την ευρωπαϊκή κουλτούρα άμυνα σε συλλογική λοιπόν εκπαίδευση, όπω την αποκαλούμε πάρα πολύ σημαντική, στο όλο αυτό πεδίο τη ε, ανάπτυξη δυνατοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ τα στρατηγία είναι ένα σημείο κλειδί γιατί είναι το επίπεδο ε, που ε, πραγματικά εργαζόμαστε στο πλαίσιο των ασκήσεων να τελειοποιήσουμε τις διαδικασίες να τις βελτιώσουμε. Ξέρετε ότι πρόσφατα επανεξετάσαμε και αναθεώρησαμε τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων ώστε να τις προσαρμόσουμε καλύτερα ε, σε αυτή την έννοια της συνολικής προσέξης και της κοινή δράσης. Και αυτό γίνεται κυρίως μέσω των ασκήσεων. Επίσης ατομική εκπαίδευση, κατάρτιση, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό βέβαια ιδιαίτερα γιατί ο Hans Μπένχαρτ ε, και το ΣΕΜ5 επίσης ε, έχουν να πούν πράγματα. Άρα κερδίζουμε χρόνο, περνάω λοιπόν αυτό το σημείο και να πω μόνο σύντομα ότι τον Οκτώβριο το Στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνοιξε ένα πάρα πολύ, ε, ε, οργάνωσε ένα ανοιχτό σεμινάριο στο οποίο προσκάλεσε και τις ευρωπαϊκούς παράγοντες και φορείς, αλλά πέραν αυτών και τα κέντρα εμπειρονομοσύνης του ΝΑΤΟ για τον τομέα πάντα της εκπαίδευσης κατάρτισης. Συμμετείχα σε αυτό το σεμινάριο λοιπόν που είχε ως θέμα τον χρόνο για βελτίωση και συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Θέλουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την όθηση, αυτή την νομή που υπάρχει για να προχωρήσουμε. Μία λέξη μόνο για την εκπαίδευση ξένων στρατευμάτων. Να πω ότι ήδη συγκεκριμένα έχουμε τεχνογνωσία τεχνογνωσία που τη βλέπουμε στη Σομαλία, στο Μάλι και περιλαμβάνεται αυτό στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ως ένα ε, στόχος μας να προωθήσουμε δηλαδή αυτό το πολύ σημαντικό μέσο και εργαλείο πρόληψης. Και βέβαια ρόλο κλειδί δεν έχει να δραματίσει πάλι εκπαίδευση. Λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα. Το στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε εντολή από τη Στρατιωτική Επιτροπή πέρυσι στο τέλος της χρονιάς να προχωρήσει σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο δράσης, ε, το οποίο εκπονείται βέβαια σε αυτή τη φάση. Στόχος μας είναι να επεξεργαστούμε τις ανάγκες μας ε, και να προβούμε και στις απαραίτητες δράσεις εκπαίδευσης κατάρτισης σε πλήρη συντονισμό και με τους άλλους φορείς και με τα κράτη-μέλη. Και με μια άλλη εργάνωση που έχουν πάρα πολλά κοινά, το ΝΑΤΟ δηλαδή. Όλοι μαζί έχουμε μια δυναμική, πραγματικά, το επίπεδο τη Επιτροπής, για να τα καταφέρουμε. Εδώ ε, θα σταματήσω. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πόρτσιο αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να σεβαστώ τα χρονικά όρια που μας θέσατε. Κατά πρώτον, να εξηγήσω κάτι. Παρόλο που το δικό μας τάγμα πρόκειται να ολοκληρώσει τη δράση της με ασκήσεις που έχουν μετακινηθεί προς το MB7 με τον κύριο Μιώτσο υπεύθυνο. Οι ασκήσεις όμως όπως είπε και ο ταξιέρχος είναι πολύ σημαντικές. Σημαντικές για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο που ε, υπάρχουν περισσότεροι πόροι. Ένα δεύτερο σημείο που είναι πολύ σημαντικό και το οποίο αφορά και τη διάσταση είναι ότι η εκπαίδευση είναι εθνική ευθύνη. Τα κράτη-μέλη έχουν πολύ ισχυρές απόψεις για τα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν το δικό μας, η δική μας δύναμη έρχεται να συμπληρώσει τα όσα ορίζει η κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προσπάθειες κυρίως των κρατών μελών. Τώρα, ποια πολιτική ακολουθούμε στην ε, κοινή πολιτική άμυνα και ασφαλεία για την εκπαίδευση. Μετά απ' όλα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει περισσότερο συντονισμένη και σφαιρικότερη προσέγγιση ώστε να μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην εκπαίδευση ε, διδάγματα από το παρελθόν, από ασκήσει που έχουν ήδη δεξιχθεί. Γι' αυτό το τμήμα των ε, διδαγμάτων είναι κάτι που και τη δική μας υπηρεσία. Δεύτερο τμήμα προσπαθειών όπου εντοπίζουμε και εμείς τη δράση μας είναι οι βέλτιστες πρακτικές και ο εντοπισμό τους. Είναι αυτό που ονομάζουμε MMA. Παρακολουθούμε δηλαδή για να δώσουμε συμβουλές. και προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης που ε, εντοπίζουμε στους διάφορους εκπαιδευτές. Όπως είπε ο κύριος Λερού, βρισκόμαστε σε δύσκολη δημοσιονομική περίοδο και πρέπει να δούμε με προσοχή τους στόχους της εκπαίδευσης. Ένα από τα βασικά τα στοιχεία που ε, μας ενδιαφέρουν ε, για την εκπαίδευση είναι να λαμβάνουμε όπως τη διάσταση του φύλου και την επιγράμμιση με τις επιταγές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι σημαντικό και κατά την διεξαγωγή των επιχειρήσεων αλλά και για την εκπαίδευση σε τρίτες χώρες. Και βεβαίως το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο είναι εξίσου σημαντικά. Θα ήθελα πολύ γρήγορα να σχολιάσω τις δράσεις που έχουμε θερισπέρα πέρα στο 2013 και το τι προγραμματίζουμε για το 2014. Έχουν γίνει προσπάθειες όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους προκειμένου να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση. Βέβαια αυτή η φράση είναι πολύ πιασάρικη αλλά πρέπει να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε για τη σφαιρική προσέγγιση. Θα μπορούσε να καλύπτει την επικοινωνία της ΕΕ της εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι πολλά άλλα πράγματα. Όμως όταν υπάρχουν 50 άνθρωποι σε μια αίθουσα, 50 διαφορετικέ απόψει θα υπάρχουν για την ε, σφαιρική προσέγγιση. Το θέμα όμω είναι να δούμε τι γίνεται όντω με την επικοινωνιακή πολιτική. Το κατά πόσο χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα, όλα τα εργαλεία που βρίσκονται στο κουτί μα. Χθε, έλεγα κάποιους ε, ανθρώπους ε, του ιδιωτικού τομέα στην εκπαίδευση ότι το κουτί εργαλείων κάποιες φορές χρειάζεται και νέες λύσεις για να μπορεί κανείς να σωματώνει και τα διδάγματα της πείρας του, το όσα έμαθε στην πράξη. Όπως θα ξέρετε, και τώρα θα αφήσω τις λεπτομέρειες στον καλό φίλο, τον Hans Bernard Weiser, η ε, εκπαίδευση στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι ε, μια πολύ σημαντική διάσταση και αυτό και θα ακούσουμε τόσο όσα κάνει στην Ελληνική Ακαδημία. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι να εκπαιδεύσουμε και το κοινό μας στο τι προσφέρουμε αλλά και αντιστρόφως δηλαδή να δημιουργούνται προγράμματα εκπαίδευσης για συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Όπως είπε ο ταξιέρχος Λερού, ε, συνεργαζόμαστε στενά και με το στρατιωτικό προσωπικό. Ο τρίτος πυλώνας των προσπαθειών που γίνονται από την Κοινή Πολιτική Ασφαλής και Άμυνας είναι η λεγόμενη PCC. Τον Οκτώβριο του 2013 οργανώθηκε για δεύτερη φορά συνάντηση των ε, επικεφαλής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στις Βρυξέλλες ήρθαν ε, ειδικοί από όλες μας τις επιχειρήσεις και αποστολές. Αυτά παράλληλα με το εργαστήρι που οργανώθηκε από την Ιγιουμπάς. Αυτό ήταν πολύ χρήσιμο από άποψη δικτύωσης πρώτα απ' όλα. Όλοι μπόρεσαν να ανταλλάξουν ε, τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους ε, και αυτά θα τροφοδοτήσουν στη συνέχεια και την εκπαίδευση, αλλά πραγματικά η δικτύωση που μπόρεσε να γίνει ήταν πολύ σημαντική, την εκτίμησαν όλοι και στο δεύτερο εξάμεινο το 2014 θα το επαναλάβουμε. Θα το επαναλάβουμε ελπίζοντας ότι θα είναι τόσο ωραίο όσο την περασμένη φορά. Υπάρχει ένα μάθημα ανώτερου κυκλού CSDP ε, της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Ο Μπέρναντ μπορεί να σας δώσει κάποια περισσότερα στοιχεία γι' αυτό και υπάρχει και ένα σεμινάριο για τα θέματα πολιτικής ασφαλείας και άμυνας που επικεντρώνεται κυρίως στην Κίνα. Η Κίνα ε, γίνεται ένας από τους πρώτους μας συνομιλητές και είναι ένα από τα σημεία που θέλουμε να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή. Η ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Έχω παρουσιάσει τα συμπεράσματά μας και σε αυτό τον τομέα με τη σχετική έκθεση που ετοιμάσαμε. Θέλουμε να υπάρχει κάποιο είδους κοινή αντίληψη για τα θέματα αυτά. Για τη διασυνοριακή μας δράση θέλουμε να καλύψουμε την ε, χαρακτήρα μας από το παρελθόν. Το ίδιο και με την ανάλυση εχθροπραξιών ή την ανάλυση ευάλωτων καταστάσεων. Τώρα, για το τι γίνεται πριν την ανάπτυξη των δυνάμεων και με το διεθνές προσωπικό, το θέμα είναι ευαίσθητο γιατί κάποια κάτι μέλη ήδη έχουν πολύ καλά μαθήματα στις δικές τους ε, ακαδημίες για την φάση πριν την ανάπτυξη. Το να δίνεται μια ευρωπαϊκή διάσταση βέβαια και μάλιστα ενός μεγέθους για όλες τις περιπτώσεις είναι κάπως περίπλοκο. Τα κάτι μέλη δεν είναι τόσο πρόθυμα να το δεχτούν. Πρέπει να βρούμε όμως έναν τρόπο να ανακουφίσουμε και τις ευρωπαϊκές ευαισθησίες σε αυτή την περίπτωση, ειδικά και αποσπασμένο προσωπικό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει και το κοινό πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ. Έχετε ακούσει πως συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΕ, ο οποίο δίνει πρόσβαση σε ένα νέο εργαλείο το οποίο ονομάζεται Goalkeeper. Τερματοφύλακα δεν είμαι φαν των ποδοσφαιρικών, αλλά θα μπορούσε να ονομάζεται και αλλιώ ε, το πρόγραμμα αυτό. Ε, πρέπει να το καταπιούμε. Τέλο πάντων είναι ένα λογισμικό που ετοιμάστηκε και ενσωματώνει όλη τη γνώση που διαθέτουμε για το τι μαθήματα προσφέρονται από τι ακαδημίες ε, λόγω χάρη για την ε, Ακαδημία, τη Στρατιωτική Ακαδημία Σαντάνα στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Μπορούμε έτσι να προσφέρουμε γνώση και σε εξωευρωπαϊκούς ενδιαφερομένους. Επίσης η συνεργασία με τον ΟΗΕ θα ετοιμαστεί έκθεση πρόοδου μέχρι τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες η έκθεση θα συνταχθεί ως το τέλος του χρόνου οπωσδήποτε. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, έχω μαζί μου τον συνάδελφο Χορς Χούκορ, ο οποίος θα μπορέσει να σας δώσει περισσότερα στοιχεία αν χρειαστεί. Επίσης υπήρξε πρόταση για ενδυνάμωση της εκπαίδευσης για την ασφαλεία και την άμυνα. Απόφαση του Συμβουλίου το 2013 μάλιστα έριξε φως στα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής που θα χρειαστούν Ξέρετε ότι η εκπαίδευση χρηματοδοτείται από, την, από τα κονδύλια για την ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και επιτόπου εκπαίδευση πέραν από την θεωρητική για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση συγκρούσεων. Ε, θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου λόγω των χρονικών περιορισμών. Η δεύτερη φάση της δράσης μας χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80%. Τα υπόλοιπα χρηματοδοτούνται από, τα, από 13 κράτη-μέλη που είναι συμβαλόμενα μέρη στο καταπίστευμα. Και το δεύτερο μέρος, όπως σας είπα, ασχολείται με θέματα της φάσης πριν την ανάπτυξη των δυνάμεων. Πολύ σύντομα. Εδώ προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το λεγόμενο IDL, την εξαποστάσεως δηλαδή, τον εξαποστάσεως χειρισμό μέσω διαδικτύου και ε, επικεντρωνόμαστε στις Βρυξέλλες αλλά θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε και περισσότερα μαθήματα. Ο ταξίρχος Λερού μίλησε για το συνδυασμό της εκπαίδευσης με τον εξοπλισμό. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας, ιδίως μάλιστα καθώς είναι ένα από τα πιο δύσκολα. Όπως γίνεται με την αναπτυξιακή βοήθεια, μερικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκπαίδευση, μπορεί στη συνέχεια να στραφούν εναντίον ε, του προμηθευτή της υπηρεσίας. Δηλαδή, στις τρίτες χώρες μπορεί ο εξοπλισμός, εάν παραμένει στα χέρια τους, να χρησιμοποιηθεί εναντίον ημών ή και άλλων ομάδων. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές που σχεδιάστηκαν το 2003 και η αντίληψη για την εκπαίδευση στην άμυνα και την ασφάλεια του 2004 έχουν γίνει λίγο απαρχιωμένες. Πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα δράσης διεπηρεσιακό, το οποίο να καλύπτει και τη CPCC και την UMS. Να προβλέψουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και να προκύψει ένας νέος κύκλος μαθημάτων που να είναι πιο προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Με συγκεκριμένο κύκλο, εκπαιδευτικό κύκλο ή διάφορους εκπαιδευτικούς κύκλους, καθώς και ένα σύστημα ε, που να είναι το κατάλληλο. Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank Θα ευχαριστώ, λέει ο κύριος Βάσερετ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσίσω το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Άμυνας. Πρόκειται για ένα κολέγιο στο οποίο προετοιμάζουμε το προσωπικό. Έχω φέρει εδώ μαζί μου και μία παρουσίαση με διαφάνειες. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να σας το δώσουμε, να έχετε και το χρόνο να το μελετήσετε. Η γραμματεία πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Όσον αφορά το κολέγιο, άμυνας της, που βρίσκεται εδώ στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι σκοπός μας είναι να προωθήσουμε όλες τις επιχειρήσεις της κοινή ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στόχους πολιτικής της κοινή εξωτερικής πολιτικής. Σκοπός μας είναι επίσης να προβάλλουμε μία στρατηγική, μία πολιτική νοοτροπία όσον αφορά την κοινή στρατηγική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, να στηρίξουμε επίσης στα πλαίσια αυτών των κοινών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες εταιρικέ σχέσεις και την συμμετοχή των κρατών μελών στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το Κολέγιο Άμυνας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου του Απριλίου 2013 έχει αποφασιστεί να λειτουργεί υπό την ε, αιγίδα της ΥΠΑ ε, εκπροσώπου και βεβαίως ενσωματώνεται στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης από κοινού με άλλους φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη λειτουργία του δικτύου, βεβαίως, υπάρχει αυτή η δομή που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, η Διευθυντική Επιτροπή με την συμμετοχή των κρατών μελών και τις αποφάσεις καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ε, αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι των ε, κολεγίων και της γραμματείας του Κολεγίου Άμυνας των Βρυξελών, έτσι, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι αυτοί στον σχεδιασμό και στις μελλοντικές δραστηριότητες του Κολεγίου. Δύο λόγια για την χρηματοδότηση. Τι προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης σε είδος όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης. Τα κράτη-μέλη μπορεί να συμμετέχουν όσον αφορά βεβαίως την δέσμευση των κρατών μελών και στο ύψος και στο βαθμό της δέσμευσής τους συμμετέχουν. Δεύτερον, στήριξη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Τρίτη δυνατότητα στήριξης χρηματοδότησης, τα κράτη-μέλη, οι βρήματα, οι άλλοι μπορούν να συνεισφέρουν για τη χρηματοδότηση κάποιου ειδικού προγράμματος ή σχεδίου και βεβαίως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου καλύπτει τα έξοδα της λειτουργίας και βλέπετε εδώ το ποσό, το συνολικό ποσό για ένα έτος είναι 535.000 ε, ευρώ. Το 60% του προϋπολογισμού ουσιαστικά διατίθεται για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες και βεβαίως υπάρχει και μία δυνατότητα συγχρηματοδότησης κάποιων ε, σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης από μέρους των κρατών μελών. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ένα μόνιμο προσωπικό 8 ατόμων και εδώ βεβαίως βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να φανεί λίγο για μόνιμο προσωπικό. Έχουμε όμως εξαιρετικά καλή συνεργασία με τους ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες, με το κέντρο της Γενέβης για την ε, πολιτική ασφάλειας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ειδικά προγράμματα κατάρτισης που οργανώνουμε από κοινού με το Ινστιτούτο αυτό. Δύο λόγια τώρα για την Εκτελεστική Επιτροπή, το Εκτελεστικό Συμβούλιο, βρίσκεται εδώ στις Βρυξέλλες. Σε ετήσια βάση γίνεται η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του κολεγίου καθώς και η παρακολούθηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων και αποστολών. Αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Και βεβαίως όλες οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας παρακολουθούνται και πολλές φορές υπάρχει και η σύσταση ειδικών επιτροπών. Δύο λόγια για τα δίκτυα και τη δομή των δικτύων. Από τότε που ιδρύθηκε το 2005 το κολέγιο έχουμε συμμετάσχει σε συνεργασία με πάνω από 60 ε, εθνικούς φορείς και Ινστιτούτα στα πλαίσια της άμυνας, της πολιτικής ασφάλειας. Όλα αυτά τα 60 Ινστιτούτα και φορείς και οργανισμοί συμμετέχουν στο δίκτυο, βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, με σκοπό βεβαίως να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ε, επιχειρήσεις και όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κοινή ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Αυτή η συνεργασία βεβαίως ενδυναμώνεται και με την συνεργασία μεταξύ της στρατιωτικής και πολιτικής πτυχής Έχουμε δηλαδή μια πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση. Όσον αφορά τώρα το εκπαιδευτικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας, βλέπετε μια πυραμίδα. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα επίπεδα και τους βαθμούς των ε, συμμετεχόντων και όλο το φάσμα των διαφορετικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων. Εδώ βλέπετε την ανάπτυξη συστημάτων τηλεεκπαίδευσης μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων. Βεβαίως έχουμε και μια σειρά προγραμμάτων που γίνονται με την συμμετοχή σε σεμινάρια και προγράμματα που όλα αυτά βεβαίως ε, λειτουργούν υπό την αιγίδα της κυρίας Άστον. Τι κάνουμε πολύ συγκεκριμένα. Στήριξη γενικότερα των επιχειρήσεων της κοινή Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, μαθήματα και σεμινάρια υψηλού επίπεδου για τους ανώτατους αξιωματικούς, αποστολές που έχουν σαν σκοπό την κατάρτιση επικεφαλής μελών των ενόπλων δυνάμεων καθώς και των γενικών επιτελείων. θεματικά προγράμματα, μία εξάπλωση διαστημική πολιτική, ασφάλεια του κυβερνοχώρου, συνεργασία εξοπλισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και εξειδίκευση προσωπικού όσον αφορά παραδείγματο χάρη κάποιες στρατηγικές αποστολές, σχεδιασμός επιχειρήσεων και ειδική στήριξη κάποιων ε, αποστολών στήριξη και συντονισμός κάποιων ειδικών αποστολών και εμπειρογνωμόνων. Από το 2008 έχουμε και προγράμματα ανταλλαγών νέων αξιωματικών. Είναι ένα σύστημα ανταλλαγών που έχει εμπνευστεί από το Εράσμος. Και αυτό βεβαίως με σκοπό να αυξηθεί ο μικτός χαρακτήρας και ο διεπιχειρησιακός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών ε, ενόπλων δυνάμεων. Αυτό στοχεύει βεβαίως κυρίως κατάρτιση αξιωματικών, ιδιαίτερα για αποστολές στα πλαίσια της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, καθότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον και μια νοοτροπία ευρωπαϊκή μεταξύ των νέων αξιωματικών. Εδώ αναφερόμαστε στις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει ακριβώς επειδή αυξάνονται οι αποστολές και οι επιχειρήσεις ασφαλείας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάποια προγράμματα που απευθύνονται για τα Δυτικά Βαλκάνια, και ένα ειδικό πρόγραμμα για την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Προγράμματα με αντικείμενο την Κίνα και το Μάρτιο του 2014 ένα πρόγραμμα ένα σεμινάριο με πολύ μεγάλη συμμετοχή κρατών ε, από την Ασία. Τι έχουμε κάνει από το 2008 μέχρι σήμερα. Είναι πολύ αξιόλογος ο απολογισμός των δραστηριοτήτων μας. Βλέπετε εδώ τον αριθμό των συμμετεχόντων, 6.500 στρατιωτικοί και μη. 6.500 λοιπόν όχι μόνο αξιωματικοί αλλά και αστυνομικοί διπλωμάτες σε προγράμματα που αφορούν την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις και σε αυτά πρέπει να σας πω ότι πρέπει να προσθέσουμε τα παρόντα προγράμματα που βρίσκονται εν τα οποία συμμετέχουν 1.200 άτομα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το υλικό που χρησιμοποιούμε για αυτά τα προγράμματα κατάρτισης και νομίζω ότι γνωρίζετε όλοι το έντυπο υλικό μας. Σας έχουμε εξάλλου δώσει κάποια από αυτά σε όλα τα μέλη της Επιτροπής για τα σεμινάρια που αποφθήνονται στο διοικητικό προσωπικό Leadership Seminars προετοιμάζουμε ένα νέο εγχειρίδιο το οποίο σας υπόσχομαι να σας το στείλω. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος πόσιο δηλαδή οι νέες αποστολές του κολεγίου που είναι η στήριξη για συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούν τη διαχείριση κρίσης στα πλαίσια των κοινών ευρωπαϊκών ε, πολιτικών ασφάλειας και άμυνας. Ιδιαίτερα αυτά απευθύνονται σε μη στρατιωτικούς και εδώ το κολέγιο έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υλικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από προσωπικό το οποίο συμμετέχει σε μη στρατιωτικές αποστολές, όπως παραδείγματο χάρη την επιχείρηση Αταλάντα, το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε παραδείγματο χάρη από τους συμμετέχοντες στο Γενικό Επιτελείο της επιχείρησης Αταλάντα. Στηρίζουμε λοιπόν και θα το κάνουμε όλο και περισσότερο και μη στρατιωτικές αποστολές στο μέλλον. Επίσης, μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μελλοντική μας δραστηριότητα κατάρτισης εδώ στις Βρυξέλλες και θα εξετάσουμε και τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα προγράμματά μας για την ανάπτυξη δυνατοτήτων και θεσμών επιτόπου σε κάποιες χώρες τις οποίες διεκπαιρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρήσεις. Βεβαίως και πολλά άλλα μπορούμε να αναπτύξουμε. Θα σταματήσω όμως την παρουσίασή μου εδώ αλλά βεβαίως αν έχετε ερωτήσεις ε, με μεγάλη χαρά θα απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τη συνεργασία με άλλους εξωτερικούς εταίρους, όπως για παράδειγμα την αμυντική ακαδημία του ΝΑΤΟ. Έχετε συνεργασία ή όχι. Και με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως βέβαια τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αλλά και το Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Κέντρο ή άλλους οργανισμούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, αλλά έχουν κάποια σχέση, Frontex, Europol. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Κύριος Γκάλερ. Attention German, ich spreche jetzt weiter auf Deutsch. Θα μιλήσω γερμανικά. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας Νομίζω κανείς δεν διαφωνεί για το πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια, πόσο αποτελεσματική είναι η δράση σας και πόσο σημαντικός είναι αυτός ο οργανισμός. Και φυσικά ξέρω ότι υπάρχει το θέμα της πρόσληψης προσωπικού, ιδιαίτερα από μέρους κρατών μελών. Ξέρουμε ότι το μη στρατιωτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ακόμα ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και ξέρω ότι σίγουρα χρειάζεται εδώ μια νέα κατάρτιση για όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιες αποστολές. Αυτό που με ξάφνιασε όταν είδα τον προϋπολογισμό σας, ότι το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού απευθύνεται στην πληρωμή των εμπειρογνωμόνων. Από μέρους δηλαδή εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που συμμετέχουν στις διάφορες επιχειρήσεις. Εμείς ξέρουμε, παραδείγματο χάρη, ότι για κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις τα γενικά έξοδα, τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται από άλλους πηγές κρυβατορός, όπως ο μηχανισμός Αθηνά. Κατάλαβα καλά ή όχι, δεν ξέρω. Έχω καταλάβει ότι όποιος συμμετέχει σε μια επιχειρήση, να σας το πω πολύ απλοϊκά, χρηματοδοτεί ως ένα βαθμό την επιχείρηση αυτή. Και όταν μιλάμε για redeployment training, δηλαδή μια κατάρτιση πριν να αναπτυχθεί και εξελιχθεί μια τέτοια αποστολή επιχείρηση, η χρηματοδότηση δεν ε, προβλέπεται εκ των προτέρων. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω καλά ή πρόκειται για άλλου είδους αποστολές με διαφορετικούς κανόνες. Επίσης, φαντάζομαι έχετε κάποια αξιολόγηση, εκτίμηση των συμμετεχόντων στα προηγούμενα σεμινάρια κατάρτισης. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο σε στρατιωτικούς, αλλά και στο υπόλοιπο προσωπικό που συμμετέχει. Πώς το εκτιμούν. Η προετοιμασία μιας αποστολής είναι κάτι που συμπεριλαμβάνει παραδείγματο χάρη και γλωσσικά θέματα. Δηλαδή, μία αποστολή σε μία γαλλόφωνη αφρικανική χώρα προϋποθέτει ότι όλοι οι συμμετέχοντες καταλαβαίνουν και μπορούν να συνεννοηθούν στη γαλλική γλώσσα. Γιατί μιλήσατε για την Ρωσία, για την Κίνα, και για άλλες χώρες. Αναρωτιέμαι όμως, εμείς έχουμε ζωτικά συμφέροντα πολύ πιο κοντά σε περιοχές όπως η Αφρική. Τα έχουμε καλύψει όλα αυτά. Δεν αναφερθήκατε πολύ, γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτά προς το παρόν. Αν απαντήσετε μπορώ να έχω και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάλερ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Ποιος θέλετε να ξεκινήσει. Let's, get this uh, another order, yeah? Εντάξει, ανάποδα αυτή τη φορά. Βάισερτ. Ευχαριστώ. Το πρώτο ερώτημα που θέσατε κύριε Πρόεδρε είχε να κάνει με την ε, Ακαδημία μας και τη συνεργασία με τέρους όπως είναι το Κολέγιο στη Ουνάτο στη Ρώμη και άλλους. Πράγματι, Έχουμε κάποια συνεργασία με το NDC. Παρέχουμε επίσης πρόσβαση στο σύστημα μελέτης εξ αποστάσεως ε, που το διαδικτυακό και επίσης ε, όταν τα μαθήματα του NDC εστιάζουν ε, στο μαθησιακό περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουμε και εμείς εκεί και έχουμε πολύ στενή συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης. Το Ινστιτούτο Στατικών Μελητών είναι πλήρες μέλος, αναφέρεται και στα καταστατικό μας. Επίσης έχουμε συνεργασία με τη ΣΕΠΟΛ, την Αστυνομική Ακαδημία δηλαδή, και συμμετέχουμε σε κοινά μαθήματα. Τα δύο τελευταία χρόνια επίσης Αναπτύξαμε κατάρτιση και στήριξη στο πλαίσιο της συνεργασίας των των εξοπλισμών με τον Οργανισμό Άμυνας. Δύο μαθήματα με τον ΕΝΤΑ, τον Οργανισμό Άμυνας. Um, we... Με το δορυφορικό κέντρο έχουμε στενή συνεργασία. Μας στέλνουν σε τακτά διαστήματα προσωπικό τους για να το εκπαιδεύσουμε και επίσης στέλνουμε μιλητέ και υλικό για το έργο του Σάτσεν. Σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες στα μαθήματα και την αποζημίωση, τα έξοδα ε, ταξιδίου και διαμονής. Ο μηχανισμός στο πλαίσιο της δικής μας Ακαδημίας έχει ως εξής. Πληρώνουν μόνοι τους οι συμμετέχοντες ε, τις δαπάνες τους, ε, αλλά ε, στην περίπτωση εισόδου, ε, το entry project δηλαδή, εκεί καταβάλλονται από εμάς τα, τα έξοδα. Σε ό,τι αφορά προαναπτυξιακή φάση, το κόστος αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να καλυφθεί από την Ένωση, από τον προβλησμό της Ένωσης, αξιολόγηση των συμμετεχόντων στα μαθήματα. Αυτό το κάνουμε για όλα μας τα μαθήματα, σε τακτά διαστήματα. Για τα μαθήματα που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ θετικά τα σχόλια. Θεωρούνται τα μαθήματα ότι είναι σημαντικά και αυτά καθευτά μαθήματα, αλλά και για την ε, εργασία έπειτα των ανθρώπων αυτών, είτε στις χώρες τους, είτε εδώ, γιατί για τη στελέχωση της ΕΕΔ ή άλλων οργανισμών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας. Και αυτά, όλα, όλοι αυτοί οι οργανισμοί εκτιμούν τη δουλειά μας. Στο πλαίσιο του έντρι γιατί του και και τη Βόρεια Αφρική για τη συμμετοχή στο μάθημα. Και σε χώρες Μεσογείου παρέχουμε πρόσβαση. Πριν από τις θερινές διακοπές είχαμε ένα μάθημα αφιερωμένο αποκλειστικά στις χώρες αυτές. Αλλά δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα στην περιοχή αυτή. Ελπίζω να κάλυψα τα ερωτήματα. Πόρτζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι. Σε ό,τι αφορά το feedback για το τι έχουμε διδαχθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια κομμάτι. Έξω σημαντικό με, το, με την κατάρτιση των μαθημάτων. Πάντα ζητάμε feedback από τις αποστολές μας. Άρα έχουμε επιτόπου λοιπόν ε, λαμβάνουμε τις πληροφορίες για να τις αξιοποιήσουμε. Διστάζω βέβαια να πάρω πολύ σοβαρά υπόψη με αυτά που λένε οι συμμετέχοντες, που λένε ότι ήταν τέλεια τα μαθήματα και τι καλός που ήταν ο ε, δάσκαλος. Το θέμα είναι όσο είναι εκεί ε, να έχουμε επαφές με τους μαθητές και με το CPCC και παίρνουμε από αυτού feedback. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά θέματα, είναι πολύ πολύπλοκο το πρόβλημα. Ακριβώ λόγω τη κατάρτιση του προπολογισμού, τη είδου του προπολογισμού. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο συνολικό προπολογισμό για τι αποστολέ ε, στο πλαίσιο τη ΚΑΠΑΠΙΑΛΦΑ από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014, 18 μήνε δηλαδή, είναι 12,3 εκατομμύρια. Ο προπολογισμό ε, για το IFS για 6 χρόνια από το 14 στο 20 είναι 2,8 δις. Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ε, κονδύ, τον προπολογισμό του μέσου του μηχανισμού σταθερότητα. Για τι ανθρωπίε των χώρων μπορούμε, αλλά όχι για, για το δικό μας προσωπικό. Πρέπει να βρούμε αλλού τα χρήματα. Και όπω έχει κατάσταση με τον προπολογισμό σήμερα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερω δύσκολα. Τέλο, σε ό,τι αφορά το γλωσσικό ζήτημα. Οι Γερμανοί που εκπαιδεύονται για να πάνε σε μια γαλλόφωνη χώρα κτλ. Ακούστε, φυσικά έχουμε το πρόβλημα με το τι γίνεται με την εκπαίδευση. Φαντάζομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις ε, η γλώσσα που μιλάμε όλοι γιατί και εγώ Ιταλό είμαι, αγγλικά μιλάω έτσι τώρα, τέλο που δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Το θέμα είναι να βρούμε τον άνθρωπο με τις κατάλληλε δεξιότητε. Τώρα ε, θα ε, χρειαστεί να μιλήσει την Καϊ Ουρντού για να πάει στη χώρα εκεί. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ε, Ταξίαρχη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για να συμπληρώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Είπατε τι κάνουμε με εξωτερικού οργανισμού. Λόγω χάρη το κέντρο δορυφόρων. Είναι ένα σημείο αναφοράς συνεχέ και διαρκέ τη ασκήσεις μα. Διαρκώ το χρησιμοποιούμε είτε σε αθλητικέ ασκήσεις, σε ασκήσει όπω η Μίλεξ, είτε άλλε που είναι στρατιωτικέ και πολιτικέ. όπως οι ασκήσει CME. Για να απαντήσω λοιπόν πιο συγκεκριμένα, για το δορυφορικό κέντρο πρόκειται για έναν συνομιλητή μόνιμο. Για την Αθηνά. Ακούστε με, κύριε Βουλευτή. Ε, νομίζω η αναθεώρηση του μηχανισμού Αθηνά φέτος είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί. Ελπίζω να τεθεί. Αλλά πραγματικά καλή τύχη για όσα εκφράσατε τόσο επιθυμία, νομίζω ότι μια διεύρυνση του μηχανισμού Αθηνά είναι μια καλή ιδέα. Και είδαμε με το πέρας του χρόνου ότι όλο αυτό μπορεί να οργανωθεί. Τώρα, οι περιορισμοί λόγω του τρόπου χρηματοδότησης, που δεν ε, αντιστοιχεί σε δημοσιονομική γραμμή μόνιμη και διακριτή, είναι κάτι που είναι ένα θέμα. Ε, επειδή δεν υπάρχει αντιστοιχεία με τις πολιτικές ε, δράσεις εδώ, πρέπει να βρεθεί μια λύση και για την Αφρική, την Αφρικανική Ένωση. Αναφερθήκατε στα μαθήματα ανώτερου κύκλου, μάλλον orientation course, ε, τα μαθήματα προσανατολισμού που αναπτύξαμε σε συνδυασμό με την, Κίνα και επίσης για το Περιφερειακό Φόρουμ ΑΖΕΑΝ. Έχουμε κάνει περισσότερα για την Ασία, είναι η αλήθεια, παρά για άλλες περιοχές του κόσμου. Δικαίως το παρατηρείται αυτό. Τώρα, για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, ακόμα δεν έχουν προβλεφθεί, δεν υπάρχει, δεν έχει οριμάσει το θέμα, αλλά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ό,τι γίνεται με την Αφρικανική Ένωση γίνεται κυρίως επί τόπου με τις αποστολές μας και με την Ινστιτουτική Επιχείρηση στην, στο Μάλι και στην Σομαλία. Για την εκπαίδευση προσώπων, το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Άμυνας και Ασφαλείας ακόμη δεν έχει μαθήματα για αυτό το θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, κύριοι, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις και την παρουσία τους. Τελευταίο μου καθήκον, να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Υποεπιτροπή προβλέπεται για τις 12 Φεβρουαρίου στις 9.30 το πρωί, στις Βρυξέλλες. Κυρίω τη κύριοι, Ευχαριστώ.